για να ξεκινήσουμε την επόμενη φάση της ε, κοινοβουλευτικής μας διάσκεψης που έχει υποδεχθεί τρομερά επιτυχής. Είχαμε καταπληκτικές συζητήσεις προηγουμένως για το μηχανισμό σταθερότητας και τώρα έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε εδώ τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Μάριου Σεντένου. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Μόλις φύγατε από την πρώτη συνεδρία στο Eurogroup και ήρθατε εδώ και πήγατε και στο ΕΚΟΦΗΝ. Και τώρα έχετε έρθει σε εμά για την ομιλία που θα εκφωνήσετε και θα έχουμε και χρόνο για ερωταπαντήσεις. Οι βουλευτές θα θέσουν ερωτήσεις και μετά θα δοθούν απαντήσεις. Παρακαλώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί νωρίτερα, να σηκώσετε απλώ το χέρι σα για να σα καταγράψουμε και θα σα δώσουμε το λόγο. Ναι, τα ταμπελάκια να σηκώσετε, αλλά δεν θα πάρουμε πολλού αγορητέ, διότι στι 3.45 πρέπει να περάσουμε στο επόμενο πάνελ και στο επόμενο θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην συμπρόεδρο, την κυρία Στογιάνοβα, τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή για του Προπολογισμού και τι Οικονομικέ Υποθέσει από την Βουλή τη Βουλγαρία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Γκουαλτιέρη. Κύριε Γκουαλτιέρη, κύριε Σεντένο. Κύριοι βουλευτές, κύριοι Ευρωβουλευτές. Είναι μεγάλη μου τιμή να συμπροεδρεύω και να συνδιευθύνω την ε, συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Ανυπομονώ και εγώ να ακούσω την ομιλία του κυρίου Σεντένου που θα μας μιλήσει για την μακροοικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης και την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. την πρώτη φορά που αναλαμβάνει την Προεδρία, η Βουλγαρία έχει δεσμευτεί να είναι ιδιαίτερα δραστήρια για να βοηθήσει στην ενίσχυση της ΟΝΕ. Κύριε Σεντέν, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε να συμμετάσχω σε αυτή την διάσκεψη στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας. Είναι η πρώτη μου παρουσία εδώ ως πρόεδρος του Eurogroup και χαίρομαι γιατί εδώ συμμετέχω σε μια εκδήλωση που συνενώνει τους εθνικούς ε, με τους ευρωβουλευτές. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Τα τελευταία λίγα χρόνια, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, ε, εφαρμόσαμε τον οικονομικό συντονισμό. Μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένα μείζον επίτευγμα και ένα καλό παράδειγμα Ευρωπαίας Πρωτοβουλίας. Διότι έχει ως αποτέλεσμα ε, βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής διαδικασίας με υπευθυνότητα. Είναι πολύπλοκη η διαδικασία στην οποία συμμετέχουν τα κράτη-μέλη και θεσμικά όργανα, αλλά μόνο έτσι μπορεί κανείς να οικοδομήσει την Ευρώπη. Με τους συναδέλφους μου εργάζομαι εντατικά για την εμβάθυνση της Ευρωζώνης, για την αναζήτηση λύσεων ώστε να καταστεί πιο ισχυρή και ανθεκτική να μπορεί να εργάζεται καλύτερα για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Ούτε μπορούμε ούτε θα ξεχάσουμε τον πολιτικό μας ρόλο. και ξέρω ότι μιλώ σε εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι έχετε συζητήσει σημαντικές πτυχές για την εμβάθυνση της ΟΝΕ νωρίτερα σήμερα και ακούστηκαν ε, διαφορετικές προοπτικές. Η προοπτική της Κομισιόν, της ΕΚΤ ε, και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι είναι κοινή η άποψη που έχουμε για τα πλονεκτήματα της ΟΝΕ και για την ανάγκη να ολοκληρωθεί. Και αυτό μας ενώνει. Σήμερα θα μιλήσω για αυτές τις προοπτικές από την ιδιότητά μου ως πρόεδρο του Eurogroup. Ε, για πολλά χρόνια εστίασα στη διαχείριση κρίσεων, μάλλον εστίασε στη διαχείριση κρίσεων και τώρα το Eurogroup στρέφει αλλού την προσοχή του στην ολοκλήρωση τη αρχιτεκτονική τη ΩΝΕ. Αυτό θεωρείται κάτι πολύ θετικό, διότι ουσιαστικά αποτελεί αναγνώριση όλων των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων που έγινε και ατομικά και συλλογικά για την αντιμετώπιση της χειρότερης κρίσης μετά τη μεγάλη ύφεση. Στη διάρκεια αυτή τη κρίση οι συμπολίτε δεν δεν έχασαν ποτέ την εμπιστοσύνη του στο ευρώ στο κοινό μας νόμισμα. Ακόμη και σε δειμνούς καιρούς το νόμισμά μας έχει συνεχίσει την πορεία του για να παγιωθεί ως ένα νόμισμα αναφορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχαμε νέα συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξη ε, σταθερή. Η Ευρώπη πλέον θεωρείται ένα κινητήριο μοχλό και μια το μηχανή ανάπτυξη. Παρά το γεγονό ότι αντιμετώπισε κραδασμού σοβαρού το 2015 και το 2016. Πράγματι, η νομισματική πολιτική με τις πρωτοβουλίες που έδωσε, με την, ποσοτική χαλάρωση, σίγουρα ήταν μια συνταγή επιτυχίας. Το θέμα όμως είναι ότι οι οι οικονομίες μας ε, ανακάμπτουν και για να ανακάμπτουν σημαίνει ότι είναι και ανθεκτικές και ίσως πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε ότι είναι. Για μένα αυτή η επίδοση της Ευρωζώνης που είναι σταθερή δείχνει ότι η ανθεκτικότητα των μελών της γίνεται μεγαλύτερη. Ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που νομίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σίγουρα το μεγαλύτερο εγχείρημα ολοκλήρωση στι τελευταίε δεκαετίε. Με εθνικέ μεταρρυθμίσει, με θεσμική καινοτομία στην Ευρώπη, έχουμε δείξει ότι είμαστε αποφασισμένοι να καταστήσουμε το κοινό νόμισμα μία μόνιμη επιτυχία. Αυτό τώρα που έχει σημασία είναι αυτή την αποφασιστικότητα να την κάνουμε πράξη. Η... Διότι το ευρώ είναι ένα μέσο προς την επίτευξη ενός σκοπού και όχι αυτός σκοπός είναι στη διάθεση των συμπολιτών μας για να βοηθήσει τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, ε, για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις μας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεγαλύτερη ενιαία αγορά του κόσμου για να αυξήσει την ανθεκτικότητα των οικονομιών μας για πιο ε, ε, ευρύ ανακατανομή του πλούτου, για να έχουμε και περισσότερες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες το ενέο αυτό νόσμα χρησιμεύει για να προωθήσει αυτό το πολιτικό εγχείρημα που φέρνει κοντά τους πολίτες των χωρών μας. Φυσικά εύκολα καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι το ευρώ και η δική μας δουλειά είναι να το κάνουμε όλο και πιο ισχυρό. Πρέπει να συνεχίσουμε να εξυγχρονίζουμε τις οικονομίες μας ώστε να μπορούν να αντέξουν σε μια επόμενη κρίση αλλά και να μπορούν να προσαρμόζονται στις αλλαγές που φέρνουν οι τεχνολογικές και δημογραφικές αλλαγέ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πολύ καλές ε, και σαφώς καθορισμένες πολιτικές σε εθνικό επίπεδο για να έχουμε βιωσιμότητα και στήριξη της ανάπτυξης. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να μεγαλώσουμε το δυναμικό μας, το αναπτυξικό δυναμικό. Υπάρχουν ε, στοιχεία πάνω στα οποία μπορούμε να βασιστούμε για να αφήσουμε πίσω μας ε, την κρίση και ό,τι κληροδότησε αυτή. Τώρα ζούμε καλούς καιρούς. Έχουμε ένα ευνοϊκό οικονομικό κλίμα και έχουμε και το χρονοδιάγραμμα που δίνει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να δράσουν όχι μόνο μεμονωμένα αλλά και συλλογικά. Αυτό που θέλω να πω ουσιαστικά είναι ότι τα κράτη-μέλη θα γίνουν πιο ανθεκτικά, θα ευημερίσουν περισσότερο αν αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις πτυχές ε, της ενιαίας αγοράς. Και έτσι έρχομαι στην έκθεση των πέντε προέδρων και σε αυτό που απεκάλεσαν ε, Financial Union, ε, την Χρηματοοικονομική Ένωση μέσα σε μια ολοκληρωμένη αγορά. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι μια τέτοια ένωση που θα περιλαμβάνει την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών είναι ένας σημαντικός ακρογωνιαίος λήθος για μια ευρύθμως λειτουργούσα οικονομική και νομισματική ένωση. Ένα ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα είναι η άλλη όψη της κοινή νομισματικής πολιτικής, γιατί χωρίς κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να αποκομίσουμε τα πλήρη ωφέλη του ενιαίου νομίσματος. Η κρίση έδειξε πόσο ευάλωτα ήταν τα κράτη. Αντέδρασαν οι τράπεζες, αντέδρασαν οι χώρες μέλη. Είχαμε έναν κατακαιρματισμό που προκάλεσε μεγάλες ενησυχίες. Όμως η κατάσταση βελτιώθηκε. Μόνο βαθμιαία όμως. Δηλαδή δεν είμαστε ακόμη στο σημείο που θα θέλαμε να ήμασταν. Υπάρχουν όμως βάσιμοι λόγοι να είμαστε και φιλόδοξοι και να προωθήσουμε αυτή τη χρηματοοικονομική ένωση και το ενθαρρυντικό σημάδι είναι ότι και οι ηγέτες μας θεωρούν την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ύψιστη προτεραιότητα. Αναμένονται συγκεκριμένε αποφάσει τον Ιούνιο. Είμαι επίση αισιόδοξο ότι θα καταστεί δυνατόν να τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα. Γιατί είναι σημαντικό. Διότι αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι ο κατακαιρματισμός ε, που αυξάνει το κόστος για όλους. Περιορίζει τις επιλογές των επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών. Δυσκολεύει τη χρηματοδότηση μιας καλής επιχείρησης. δυσκολεύει ε, το να βρει κανείς μια καλή ασφάλεια. Εγώ μιλάω για τον Ιούνιο, αλλά δεν το εννοώ σε ένα οδικό χάρτη. Λέω ότι απλά πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Οι συζητήσει για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης περιστρέφονται γύρω από την ισορροπία και την αλληλουχία τη μείωση κινδύνων και του επιμερισμού κινδύνων. Πετύχαμε πολλά τα χρόνια της κρίσης σε ό,τι αφορά τη μείωση των κινδύνων. Η διατέλεσα Υπουργό Οικονομικών στην Πορτογαλία και το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Διορθώσαμε τις ε, ανισορροπίες και τώρα έχουμε εμπορικό πλεόνασμα. Το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι σχεδόν 1%. Σημείωσε μεγάλη πτώση. Επίσης, ε, διορθώσαμε το τραπεζικό σύστημα, προβήκαμε σε ανακεφαλαιοποίηση των ε, τραπεζών και έχουμε νοδικές τάσεις, ε, μειώνεται και η ανεργία. Βέβαια, κάθε κρίση έχει το τίμημά τη. Έχουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά αυτά μειώνονται και το ίδιο και το δημόσιο χρέο. Με άλλα λόγια, τα του οίκου μας τα κρατούμε σε τάξη. Έχουμε αντλήσει τα διδάγματά μας από την κρίση. Βλέποντας ε, τα επίπεδα ε, του επιμερισμού ε, δημόσιο και ιδιωτικού χρέους σε σχέση χάρη με τη ΣΥΠΑ, μου φαίνεται ξεκάθαρο ότι είμαστε πίσω και έχουμε να ανακτήσουμε κάποιο έδαφος. Ο των κινδύνων είναι ένα σημαντικό ζήτημα λόγω του ότι μπορεί να επηρεάσει ε, την οικονομική κατάσταση των περιφερειών ε, και να αυξήσει την ανθεκτικότητα σε περίπτωση περίοδων ε, ισχνών αγελάδων, αν μπορώ να το πω έτσι. Η Ευρωζώνη είναι ακόμα πίσω από τη ΣΥΠΑ στον τομέα αυτό. Πρέπει και ο ιδιωτικός τομέας να μπει στο παιχνίδι για τον επιμερισμό κινδύνων θα προχωρήσουμε τους επόμενους μήνες σε αυτό το δρόμο. Δεν είναι μία ανυπέρβλητη πρόκληση. Γιατί δεν ξεκινάμε και από το μηδέν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επιφορτιστεί με την ε, τραπεζική εποπτεία και έχουμε κανόνες ε, που επιβάλλουν ε, τους πιστωτές των τραπεζών που έχουν πτωχεύσει να πληρώσουν το λογαριασμό. Επίσης, για τη μείωση των κινδύνων έχουμε ισχυρότερους τραπεζικούς ισολογισμούς με αύξηση κεφαλαίου, μείωση ε, του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όταν λοιπόν φτάσουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι από κοινού που βρισκόμαστε σήμερα, θα είναι πιο εύκολο να συμφωνήσουμε για τις ε, ε μετατροπές που πρέπει να γίνουν. Σας διαβεβαιώ ότι όλες τις ανησυχίες ε, που εκφράζονται για τον υπηρεσμό των κινδύνων τι παίρνω πολύ σοβαρά υπόψη και θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Κανείς δεν ζητά μόνιμες πιστώσεις ε, ή σκέφτεται να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο θα το εκμεταλλεύονται κάποιοι, αν μπορώ να του πω, ελεύθερους καβαλάριδες. Θέλουμε να υπάρχει ένα ανθεκτικό κίνημα με το λεγόμενο risk pooling, τη συγκέντρωση κινδύνων που έχει να κάνει και με τα ζητήματα των αντασφαλίσεων βέβαια, όχι μόνο της, του επιμερισμού κινδύνου. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τον οδικό χάρτη του Συμβουλίου του 2016 σε ό,τι αφορά τις διάφορες πτυχές της Τραπεζικής Ένωσης και δύο είναι τα βασικά σημεία. Όπως και στις περισσότερες ομισματικές ενώσεις θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Με ένα τέτοιο σύστημα θα βελτιωθεί η προστασία των αποταμιευτών, θα μειωθούν οι κίνδυνοι ενός bank run και βέβαια ο στόχος είναι γρήγορα να δημιουργηθεί και αυτός ο μηχανισμός ασφαλείας, backstop, για το νέο Ταμείο Εξυγένσης. Θα ήθελα και πάλι να κάνω μια σύγκριση με τη ΣΥΠΑ, όπου εκεί παρέχεται από το, στο, στο FDIC από τα δημόσια ταμεία αυτό το backstop ε, από το Υπουργείο Οικονομικών. Και σίγουρα θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε την πιο καλή δυνατή ο ναι. Και έρχομαι στο δεύτερο κομμάτι, την Ένωση κεφαλαίου Αγορών, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της ενίας αγοράς. Βοηθά από και δανειστές ε, να έρθουν πιο κοντά κατά κάποιο τρόπο και να βρουν τη χρηματοδότηση εκεί που την χρειάζονται. Αυτό σημαίνει επενδύσεις, ε, σημαίνει καινοτομία και αυξάνει το συνολικό μας δυναμικό ε, ανάπτυξη. διότι αν η χρηματοδότηση πάει ε, σε σχέδια βιώσιμα διακρατικά. Επίσης, η Ένωση Κεφαλαίου μπορεί να μειώσει την μεβολική εξάρτηση από τον τραπεζικό δανεισμό. Αν έχουμε λοιπόν μία ενίωση κεφάλαια αγορών θα έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα. φέρνει πάρα πολύ από τα αποτελέσματα και στι επιχειρήσει και στου πολίτε αυτό το εγχείρημα. Οι πολίτε τη Ευρώπη θα ωφεληθούν από υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξη, από περισσότερε θέσει εργασία. θα μπορέσουν να διαφοροποιηθούν και να έχουν και καλύτερε επιδόσεις ε, στι οικονομίε του Ένωση κεφαλαιών σίγουρα είναι ένα project που απαιτεί δράση σε πολλά μέτωπα. Παραδείγματο χάρη, να έχουμε καλύτερη πρόσβαση και εποπτεία των ε, κεφαλαιακών ορών πρέπει να έχουμε την κατάλληλη αρχιτεκτονική γι' αυτό. Θα πρέπει επίση τα δυσυνοριακά εμπόδια στι ζωέ αυτέ να τα άρουμε. Υπάρχουν κάποια προβλήματα όπως ασύμμετρη πληροφόρηση, θέματα αφαιρεγγιότητας, ε, η ποιότητα των ε, εγχώριων φορέων. Ε, όλα αυτά είναι δύσκολα, πολύπλοκα, αλλά σίγουρα αξίζει να τους δοθεί μια νέα όθηση και θα πρέπει αυτά τα θέματα να μπουν πιο ψηλά ε, στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν και άλλε συνέπειε που πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μα μεταξύ Τραπεζική Ένωση και Ένωση Αγορών Όσο πιο γρήγορα έχουμε πρόοδο στου δύο αυτού τομεί, τόσο πιο εύκολα θα μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφο σε άλλα σημαντικά ζητήματα, όπω είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα, κοινή δημοσιονομική ικανότητα και καλύτερων δημοσιονομικών κανόνων. Πιστεύω ότι ε, αν βρούμε τη σωστή ε, ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής αλληλεγγύης και δημοσιονομικής ευθύνης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει στη διάθεσή της ένα μηχανισμό ε, που θα συνδυάζει τα σταθεροποιητικά χαρακτηριστικά των κεντρικών προϋπολογισμών άλλων όμοιρων, ό, όριμων νομισματικών ενώσεων. Και θα επιτρέψει την ανακούφιση των χωρών που βρίσκονται σε μακροχρόνια περίοδο ύφεσης. Επίσης θα υποστηρίξει και την ε, υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής ε, της ΕΚΤ. Έχουμε πολλά αρχικά, το, το ναι, ΕΚΤ, έκθεση των πέντε προέδρων, ε, δικός χάρτης κτλ. Αυτά όμως δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίζουν και όταν είχα υποβάλει υποψηφότητα για τη θέση του Προέδρου του Eurogroup, είχα πει ότι εμεί είμαστε πολιτικοί αξιωματούχοι και ευθύνη μα και καθήκον μα είναι να εξηγούμε στου πολίτε τι μεταρρυθμίσει θέλουμε να εφαρμόσουμε. Όταν λοιπόν μιλούμε για κεφάλαιο αγορών, πρέπει να εξηγήσουμε τι εννοούμε. Δηλαδή ότι διευκολύνουμε τι νοφεί επιχειρήσει τη Φιλανδία, για παράδειγμα, να βρουν χρηματοδότηση στη Γαλλία. Ή για έναν Ιρλανδό συνταξιούχο να μπορεί να βάλει τι οικονομίε του στη Γερμανία. Μία μέσα επιχείρηση από την Ισπανία να μπορεί ε, να συγκεντρώσει κεφάλαιο στην Ολλανδία. Μιλάμε για σταδιακό άνοιγμα, για περισσότερε ευκαιρίε προ του πολίτε και προ τι επιχειρήσει. Έτσι θα εκμεταλλευτούμε το αναπτυξιακό μας δυναμικό και έρχομαι έτσι στο τελευταίο μου σημείο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία εμβάθυνσης της ΩΝΕ συμβαδίζει με τη δημοκρατική λογοδοσία και έλεγχο. Αυτό δεν θέλουμε να γίνει μόνο για λόγους βιτρίνας. Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξαν ότι υπάρχει στήριξη για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και το ευρώ. Και το ε, αποδεικνύουν αυτό και τα γκάλωπ της κοινή γνώμη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όμω να δώσουμε αυτά αποτελέσματα, να είμαστε πραγματιστέ στις λύσεις που προτείνουμε, όπω και στη διάρκεια τη κρίση, αλλά αυτό όχι ει βάρο των ε, δημοκρατικών διευθετήσεων. Οι απαιτήσει τη συνθήκη και οι νομικέ απαιτήσει θα γίνουν σεβαστέ. Δεν θα πρέπει όμω να μα παρεμποδίσουν από το να βρούμε ε, τις ε, κατάλληλες για να καλύψουμε τι προσδοκίες των πολιτών. Οι διακοινοβουλευτικές συνελεύσεις όπως η σημερινή είναι πολύ καλά παραδείγματα της αφοσίωσής μας στο να συνεχίσουμε την κοινή μα προσπάθεια για δημοκρατικές πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε Σεντένου. Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας. Έχουμε έξι αγορητές που έχουν ζητήσει το λόγο και επειδή έχουμε μόνο 18 λεπτά θα είμαστε αυστηρότατοι στο όριο ομιλίας του καθενός. Δύο ανά ομιλητή. Ο κύριος Βέρτ από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα πολύ σύντομο ερώτημα. Κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, μα είπατε ότι είμαστε σε φάση ανάπτυξη. Και πράγματι αυτό είναι αληθέ. Οι περισσότερε χώρε γνωρίζουν υψηλή ανάπτυξη και η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να καλύπτει το χαμένο έδαφο για να φτάσει στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Ωστόσο, πάντοτε υπάρχει κίνδυνο πίσω από κάθε ανάπτυξη. Θα μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι κίνδυνοι που έχετε αναγνωρίσει σήμερα. Υπερεκτίμηση των στοιχείων ανεργητικού, υπερχρέωση, διάφορες μεταβλητές που αλλάζουν από χώρα σε χώρα, είτε πρόκειται ε, για δημόσιο χρέος, είτε πρόκειται για ιδιωτικό χρέος. Θέση της ψηφιακής οικονομίας με τα μονοπόλια που μπορεί να υπάρχουν εκεί. Ε, Θεσμική κίνδυνη επίσης γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε τις ενώσεις που, για τις οποίες αναφερθήκατε, ε, την, Τελωνιακή, την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση την Κεφαλαιακή, των αγορών κεφαλαίου. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι κυρίως που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη στην Ευρώπη και η ανάπτυξη στις χώρες του ευρώ. Ευχαριστώ κύριο Σίλβα Περέιρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω το Μάριου Σαντένου η επιλογή του ως πρόεδρο του Eurogroup είναι ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον της Ευρωζώνης και για την αναθέρμανση των φιλοδοξιών για σύγκληση και ανάκαμψη του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Είναι πολύ απαιτητικό ο ρόλο που ανέλαβε, ιδίω επειδή από τον θετινό Ιούνιο δεν θα υπάρχει απλώς ένας οδικός χάρτης, αλλά ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων δράσεων για την ε, αναδιάρθρωση της Ευρωζώνης, τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης. Θέλω να κάνω τις εξής δύο ερωτήσεις. Πρώτον, στην ε, μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, τι ρόλο θα πρέπει να προβλέψουμε για την δημοσιονομική της δυνατότητα. Είστε ε, αισιόδοξο ως προς την σχέση της συζήτηση αυτής ε, και σε συνδυασμό με το Πουδουπού, με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, διότι εάν δεν συνδυαστούν αυτά τα δύο, ε, δεν θα είμαστε πολύ αξιόπιστοι ως προς τη δημοσιονομική δυνατότητα της Ευρωζώνης. Και το δεύτερο έχει να κάνει με κάτι που αναφέρατε στην ομιλία σας, τη σημασία του να διασφαλίσουμε την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της οικονομικής διακυβέρνησης και της δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Δηλαδή, από αυτήν την άποψη, η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου σε όλα τα βήματα, του Ευρω... τα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πώς σας φαίνεται, δεν θα ήταν ένας τρόπος να εγγυηθούμε την δημοκρατική νομιμοποίηση των ε, αποφάσεων της οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φίρτε από το Ουγγρικό Κοινοβουλίο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τα σχόλιά μου απευθύνονται στους επόμενους ομιλητές. Θα ήθελα να ξαναπάρω το λόγο αργότερα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χωσέ Μανουέλ Φερνάντεθ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ήθελα να χαιρετήσω τον Πρόεδρο του Eurogroup και να το ευχηθώ καλή τύχη στο ρόλο του. Είμαι βέβαιος για την επιτυχία. Επιτυχία που αν είναι επιτυχία του Πρόεδρου του Eurogroup θα είναι και επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την επόμενη Πέμπτη θα ψηφίσουμε για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τι δημοσιονομικέ προοπτικέ για του ιδίου πόρου. Συμφωνούμε όλοι ότι με την ενίσχυση τη Ευρωζώνη και τη βοήθεια των κρατών μελών που θέλουν να προσχωρήσουν, μπορούμε να καθορίσουμε μια γραμμή για το ευρώ. Και για όσους είναι μέσα και για όσους θέλουν να έρθουν μέσα. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε το backstop για την Τραπεζική Ένωση και ένα μέλλον για την Ευρωζώνη, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το, ε, τους ασυμμετρικούς κινδύνους και κραδασμούς και όσους είναι συμμετρικοί. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι απλή και συγκεκριμένη. Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα κέρδη της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως βάσει των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήταν ε, πολύ μεγάλη βοήθεια. Η ερώτησή μου λοιπόν προς τον πρόεδρο του Eurogroup είναι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να ενισχύσουμε τον προπολογισμό, διότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα ε, επιβαρύνουμε πλέον τους φορολογουμένους. Θα έχουμε ένα μεγάλο μέρος των ιδίων πόρων για να λειτουργήσει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, Ευχαριστούμε η κυρία... Η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ κύριε Σεντένου να σας καλωσορίσω στο σώμα αυτό και να σας ευχηθώ καλή τύχη. Μας παρουσιάσατε τις προτάσεις σας για το δικό χάρτη, το χάρτη πορείας για τους ερχόμενους μήνες. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κάποια σημεία που παραμένουν σαφή για την παρουσίασή σας. Στην παρουσίασή σας, το θέμα των κρατικών χρεών και το θέμα των εμπορικών ισοζυγίων. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν εάν έχετε πρόγραμμα, πρόπτικη, για ένα τρόπο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του χρέους με τρόπο πολυμερή. Και τι θα γίνει με χώρες που έχουν συστηματικά πλεόνασμα, όπως είναι η Γερμανία. Ευχαριστούμε ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, ε, ε, ευχές από πλευράς μας για καλή επιτυχία. Ε, για την Πορτογαλία που μιλήσατε, να θυμίσουμε ότι παρά την πίεση και το διαρκή εκβιασμό των ε, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπόρεσε να ξεκινήσει μια πορεία προς την ανατοποθέτηση στο σωστή πορεία και ανάκτηση κάποιων δικαιωμάτων. Να βελτιωθούν λίγο οι συνθήκες διαβίωσης ε, παρά την ε, οικονομική εγκατάλειψη της χώρας. Εδώ λοιπόν οι κανόνες της Ευρωζώνης και της ΟΝΕ ήταν μια πραγματικότητα που απετέλεσε πραγματική ε, τροχοπέδη για να προχωρήσει στην πορεία της η Πορτογαλία. Οι κανόνες και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν δεν αντιμετώπισαν το διαρκές έλλειμμα της χώρας, το δημόσιο χρέος και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η εμβάθυνση της ΟΝΕ θα σημάνει ακόμα περισσότερη εμβάθυνση αυτού του είδους των προβλημάτων και των δεσμεύσεων των τροχοπεδών. 16 χρόνια, 16 χρόνια ε, συστηματικής απόκλησης είχαμε στην περίπτωση της Πορτογαλίας και δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Ήθελα λοιπόν να θέσω ένα ερώτημα για το χρέος. Το ίδιο το χρέος των περιφερειακών οικονομιών είναι αποτέλεσμα της υιοθέτησης του ευρώ και της ΟΝΕ. Η εξυπηρέτηση του χρέους και οι ρυθμοί αντιμετώπισης και μείωσης που επιβλήθηκαν ε, οδηγούν σε γιγαντιαία παράκαμψη σε σχέση με την πορεία που θα πρέπει να ακολουθούν οι χώρε για να ανακάμψουν. Εδώ έχετε πει κάποιε φορέ ότι το πρόβλημα του χρέου στην Πορτογαλία και στι άλλε περιφερειακέ οικονομίε θα έπρεπε να επιληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, η ερώτησή μου είναι, με τι συγκεκριμένε προτάσει σκέφτεστε να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα, Ποιε είναι οι προτάσει σα για περιορισμό του χρέου, ε, ποια μέτρα θα αναλυφθούν ώστε τα πρωτογενή πλεονάσματα που χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν ακριβώς τα χρέη συστηματικά, πώς θα χρησιμοποιηθούν για χώρες που αυτή τη στιγμή μας έχουν βάλει στο φαύλο κύκλο της διαρκούς εξυπηρέτησης του χρέους. Πώς θα τα αντιμετωπίσει αυτά η εμπάθηση της ΟΝΕ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε Σεντένου. Ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας. Θα ήθελα καταρχάς να απαντήσω στις πρώτες ερωτήσεις που δέχθηκα για τους κινδύνους που συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε, που έχουμε ενώπιόν μας. Ποιοι κίνδυνοι είναι αυτοί. Εν μέρη έγκυται ε, σε, στο εξωτερικό επίπεδο, είναι εξωτερική κίνδυνη δηλαδή και πρέπει να είμαστε ενήμεροι και να είμαστε προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούμε όποτε και αν τυχόν επέλθουν. Και υπάρχουν και κίνδυνοι που βρίσκονται στο, και απορρέουν από την κρίση ακόμα. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να τους αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Ο βασικός κίνδυνος που βλέπω σήμερα είναι ο κίνδυνος της μη δράσης. Εάν δεν μεταρρυθμίσουμε περισσότερο τη ζώνη του ευρώ για να γίνει πιο ανθεκτική, πιο ικανή να αντιμετωπίσει την επόμενη κρίση, τότε δεν θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και αυτό σημαίνει φυσικά ότι Πρέπει να αντιμετωπίσουμε κινδύνους που μας έχουν κληροδοτηθεί και εξωτερικούς κινδύνους. Ο οδικός χάρτης που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ λεπτομερής ως προς αυτά τα θέματα και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε να πορευόμαστε με βάση ακριβώς αυτόν τον οδικό χάρτη, χωρίς αποκλήσεις, τότε θα καταστήσουμε την οικονομική και νομισματική μας ένωση περισσότερο ικανή να αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους. Εάν μου επιτρέπετε, θα συνεχίσω να απαντώ ε, στη μητρική μου, τα πορτογαλικά, για να πω ότι η δημοσιονομική πόρη της Ένωσης, η δημοσιονομική δυνατότητα και το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια χρηστή διαχείριση των πόρων στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ε, παράγοντες που θα κρίνουν την ε, υλοποίηση, την εξακολούθηση όλων των κοινών πολιτικών που έχουμε σχεδιάσει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάξουμε ε, το πλαίσιο όλων των ε, δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων για να τις προσαρμόσουμε στους βασικούς μας στόχους. Δηλαδή, για άλλη μια φορά. Για να γίνουμε πιο ανθεκτικοί και εμείς και η νομισματική, Οικονομική και Νομισματική Ένωση η όλη κουβέντα για τη δημοσιονομική δυνατότητα και την ενίσχυσή της είναι ιδιαίτερα εύστοχη. Πρόκειται για ένα θέμα, ένα ζήτημα που είναι τόσο πιο εύστοχο όσο ε, φαίνεται ότι εμείς αυτές τις δημοσιονομικές δυνατότητες πρέπει να τις θέσουμε στην υπηρεσία αντιμετώπισης των ασυμμετρικών κραβασμών και σοκ και στις δυνατότητες της επενδυτικές των διάφορων οικονομιών όπως εξελίσσονται στον κύκλο των ε, οικονομικών φάσεων. Αυτή λοιπόν η δημοσιονομική δυνατότητα και ενίσχυσή της είναι μια διάσταση που δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Προφανώς και αυτό ήταν μια από τις αδρές γραμμές της αρχικής μου παρέμβασης, η συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου σε όλη αυτή την ε, εξέταση, τον στοχασμό, είναι απαραίτητη. Δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε τη συμμετοχή σας και το ότι οι συζητήσεις αυτές μόνο να ωφεληθούν μπορούν από τη δική σας συμμετοχή. Τώρα για τα κέρδη της ε, ΕΚΤ είναι ευρωπαϊκή πόροι, ως τέτοιοι πρέπει να γίνονται αντιληπτοί σε τέτοιες συζητήσεις και βεβαίως το Συμβούλιο θα ε, δει συνολικά το θέμα, τις ε, δυνατότητες που προσφέρονται. Προσωπικώς είμαι υπέρ της άποψης ότι τα κέρδη αυτά είναι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να διατίθενται κατά τον ε, καλύτερο δυνατό τρόπο ε, για το σύνολο των πολιτικών μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα η Ευρωζώνη έχει σοβαρά πλεονάσματα. Πλεονάσματα που μπορεί να είναι στη μορφή των, ε, των αποταμιεύσεων συνολικά και οι μεταρρυθμίσεις που περιέγραψα της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης των Κεφαλαίων Αγορών είναι άκρος σημαντικές για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα κονδύλια, αυτοί οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν υπέρ και προς όφελος των πολιτών της Ευρωζώνης. Ο κατακαιρματισμός των αγορών η δυσκολία ή αποταμιεύσεις ε, να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για ε, επενδύσεις δημιουργούν δυσκολίες στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προβλέπονται συγκεκριμένε συστάσεις ε, μέσα από την ειδική αξιολόγηση που γίνεται για το πώς τα πλεονάσματα αυτά μπορούν να ανακατανεμηθούν και πώς η έλλειψη ισορροπίας μπορεί να ε, βελτιωθεί ε, στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Ήθελα σήμερα να μην ξεχνάμε τη σημασία των μεταρρυθμίσεων που έχουμε μπροστά μας. Διότι και αυτές θα συμβάλλουν στην καλύτερη αναδιανομή αυτών των ε, πλεονασμάτων και την καλύτερη ανάληψη από πλευρά τη Ευρωζώνη τη δυνατότητα που τη προσφέρεται από αυτά τα πλεονάσματα. Αυτό μπορεί να στηρίξει το εύρωστο της ανάκαμψης στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, αν βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας, δίνεται και ένα θετικό μήνυμα σε σχέση με τα πλεονάσματα. Ως προς το χρέος, τις σχετικές ερωτήσεις που θέσατε. Πολύ συζητημένο θέμα, ως προς το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η κρίση, έχουμε μηχανισμούς στήριξης για τη διαχείριση αυτή τη στιγμή, πολύ πιο αποτελεσματικούς από ότι στην ανάδυση αυτής της κρίσης, στο ξέσπασμα, το μηχανισμό σταθερότητας, που είναι ένα σχετικό παράδειγμα, αλλά πρέπει να εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε αυτόν τον μηχανισμό σταθερότητας για να προσαρμοστεί στις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν και που ήδη έχουμε προβλέψει. Για άλλη μια φορά πρόκειται για προσαρμογή των υπαρχόνων πόρων στη βέλτιστη δυνατή χρήση τους και ταυτόχρονα το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που, έχουμε, που εξετάζουμε τώρα θα βελτιώσουν το μηχανισμό και την όλη του εφαρμογή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον Μάριο Σεντένου και σας ευχαριστούμε για την ξεκάθαρη αυτή σας ε, δέσμευση και υπόσχεση να χρησιμοποιήσουμε αυτή την θηρίδα ευκαιρίας για να ολοκληρωθεί η τραπεζική μας ένωση και η ΟΝΕ μαζί με την ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας, την διαφάνεια και πραγματικά ανυπομονούμε για την καλή συνεργασία μεταξύ Eurogroup, Ευρωκοινοβουλίου και για τον ενισχυμένο διάλογο μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωκοινοβουλίου καθώς είμαστε συνοδοιπόροι και χτίζουμε μαζί τα θεμέλια της δημοκρατικής εκπροσώπησης στην Ευρώπη. Αυτή η διάσκεψη νομίζω ότι ακριβώς συμβάλλει στην ενίσχυση του ε, διακοινοβουλευτικού διαλόγου εν ώψη της ενίσχυσης και της ΟΝΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ τον Μάριο Σεντένου και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο τμήμα ε, της συνόδου μας. Το χρήμα για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Χαίρομαι γιατί έχω την ευκαιρία να σας απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό επί τη, επί ευκαιρία αυτής της τελευταίας καταληκτικής συνεδρίας της σημερινής ημερίδας συνεδρία η οποία θα αφιερωθεί ουσιαστικά στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο ελπίζουμε όλοι θα προσδώσει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα μέσα, τα κατάλληλα για να προετοιμάσει καλύτερα το κοινό μέλλον όλων μας. Να χαιρετήσω την κυρία Στανιάνοβα, πρόεδρο της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προϋπολογισμού και Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης της Βουλγαρίας, που θα προεδρεύσει στο πρώτο πάνελ των ομιλητών. Έχετε αυτά τα καρτελάκια που ε, θα πρέπει να αναδείξετε αν θέλετε να πάρετε το λόγο και αν θέλετε να ζητήσετε το λόγο και θα έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας. Να δώσετε λοιπόν τα καρτελάκια αυτά στους κλητήρες για να ζητήσετε το λόγο. Και χωρίς να καθυστερήσουμε περαιτέρω, προτείνω να ακούσουμε τον Επίτροπο κύριο Γκίντερ Έτιγκερ, ο οποίος βρίσκεται εδώ μαζί μας και τον ευχαριστώ. Ε, δεν μπορεί να μείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γι' αυτό είναι καλύτερο να του δώσουμε πρώτα εκείνου το λόγο. Παρακαλώ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, αξιότιμοι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω που διοργανώσατε αυτή στις δύο ημερίδες εργασίας ε, στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω μαζί σας για το μέλλον της Ευρώπης και για το μέλλον των οικονομικών της Ευρώπης. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν τρία εργαλεία πολιτικής. Κανονισμοί, νόμοι, πρότυπα, αφενός κατά δεύτερον μια πιστική επικοινωνία και κατά τρίτον η χρηματοδότηση προγραμμάτων και σχεδίων, χρηματοοικονομική δηλαδή πτυχή από τους ε, κρατικούς προϋπολογισμούς. Εμείς αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε ένα επταετές πολιετές ε, δημοσιονομικό από το 2021 και μετά. Στις 2 Μαΐου φέτος θα το καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο Επομένως, ε, μπορείτε με αυτές τις ημερίδες που οργανώνετε να δώσετε πολύ επικοδομητικές ε, συνεισφορές και ιδέες. Διότι εσείς και τα εθνικά σας κοινοβούλια είστε αρμόδιοι για τον εθνικό προπολογισμό και θα χρειαστεί πλειοψηφία για την έγκριση προπολογισμού. Είτε είναι μία ε, η Βουλή είτε είναι δύο. Αλλά η αρχή της πλειοψηφίας ισχύει παντού και για ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στην περίπτωση αυτή απαιτείται πλειοψηφία εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής Προπολογισμών, Αρτουή, βουλευτές, ε, μέλη της Επιτροπής Προπολογισμών, αλλά και όλοι οι άλλοι βουλευτές είναι αρμόδιοι για την έγκριση του προπολογισμού που φυσικά θα πρέπει να γίνει δεκτός ομοφόνος από το Συμβούλιο. Σκεφτείτε στο κοινοβούλιο σας ε, για την δημοσιονομική πολιτική της χώρας ε, να χρειαζόταν ομοφωνία. Καλή τύχη θα σας έλεγα. Εδώ χρειάζονται 27 Υπουργοί Οικονομικών. 27 Υπουργοί Εξωτερικών, Γενικών Υποθέσεων κτλ. Ουσιαστικά χρειάζονται 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Και όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Εσάς δηλαδή σας χρειαζόμαστε γι' αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο από την εκλογή Πάπα μετά από αυτά που σας είπα. Έχω πάει σε πρωτεύουσε, έχω μιλήσει με υπουργού, έχω μιλήσει με βουλευτές και θα συνεχίσω να το κάνω. Εμείς θέλουμε να έχουμε να παρουσιάσουμε ένα πακέτο, μια δέσμη μέτρων που μπορεί να είναι ικανοποιητικό για όλους. Το θέμα είναι όμως εσείς τι προσδοκάτε και τι προσδοκούν οι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Πέμπτη και την Παρασκευή υπάρχει συνάντηση των 27 πλέον σύντομα ε, κρατών μελών και δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα και καμία πρόταση δεν έχει κατατεθεί των προτέρων. Έχουμε, αν θέλετε, έναν κατάλογο, ένα μενού ε, στην επικοινωνία μας και θέλουμε να μας πείτε εσείς τι θα παραγγέλνατε, τι θα θέλατε από αυτό το μενού για την ε, Ευρώπη, για το μέλλον της Ευρώπης ε, και φαντάζομαι ότι αυτό που θα θέλατε θα ήταν προγράμματα, θέματα, εξελίξεις όπου για τον πολίτη θα υπάρχει προστιθέμενη αξία που θα είναι φθηνότερο, θα μπορεί να το χρηματοδοτήσει ε, η Ένωση αυτό το πρόγραμμα και με το οποίο πρόγραμμα θα μπορούν να λυθούν καλύτερα τα προβλήματα. Έχουμε το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο με τα παραδοσιακά του προγράμματα. Έχουμε την πολιτική συνοχής, έχουμε την κοινή γεωργική πολιτική ή το Connecting Europe δηλαδή ε, για τις οδικές ε, και σιδεροδρομικές μεταφορές για την ενέργεια ε, τα προγράμματα. Έχουμε και το Erasmus Plus για εκατομμύρια νέους που θέλουν να βιώσουν την Ευρώπη, που μετακινούνται, που συνδυάζουν, μάλλον που, δεσ... που συνδυάζουν την Ευρώπη με την κινητικότητα. Και έχουμε και το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης Αυτά είναι τα προγράμματα που έχουμε τώρα, τα παραδοσιακά. Αλλά τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν απρόβλεπτα νέα καθήκοντα και δαπάνες, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε για παράδειγμα τη μεταναστευτική, την προσφυγική κρίση, την τρομοκρατική απειλή, τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας και εξωτερικής ασφάλειας. Και ακριβώς αυτούς τους νέους τομείς η Ευρώπη δημιουργεί προσθέμενη αξία. Μπορούμε δηλαδή να εργαστούμε πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτά τα θέματα. Ήμουν στη διάσκεψη ασφάλειας του Μονάχου την προηγούμενη εβδομάδα όπου συμμετείχαν πάνω από 100 Υπουργοί Εξωτερικών και Υπουργοί Άμυνας. Και ήταν πολύ σαφές τι αναμένουν όλοι. Να μπορεί να πάρει στα χέρια της Ευρώπη την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια και να μην βασίζεται μόνο στους Αμερικανούς. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει το δρόμο προς μια αμυντική ένωση. Επίσης από κοινού ε, έχουμε αυτά τα αμυντικά προγράμματα έρευνας. Έρευνα στη βιομηχανία, πάντα για την αμυντική βιομηχανία. Επενδύουμε στην αμυντική βιομηχανία και στην έρευνα γιατί θεωρούμε ότι έχει προσθέμενη αξία ξεκάθαρα. Ένα δεύτερο παράδειγμα Πολλοί Υπουργοί Οικονομικών, Εθνικοί Υπουργοί λένε ότι η έλεγχη εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης είναι απαραίτητη μόνο εάν δεν λειτουργούν σωστά οι εξωτερικοί έλεγχοι, έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα. Όταν έχουμε δηλαδή κάποιους πρόσφυγες που φεύγουν από εμφύλους πολέμους, όταν έχουμε τούντες άσυλο, όταν έχουμε να κάνουμε με οικογενειακή επανένωση. Εγώ νομίζω ότι ελευθερία μετακίνησης και κανένας έλεγχος μεταξύ Γερμανίας, Δανίας, Σλοβενίας, Αυστρίας είναι ένα σημαντικό μεν ε, πλεονέκτημα για τον κόσμο εργασίας και για τον πληθυσμό. Αλλά είναι και μεγάλη πρόκληση. Πρέπει να βοηθήσουμε όμως και τους Βούλγαρους φίλους, τους Έλληνες φίλους, τους Ιταλούς φίλους τους φίλους μας στη Μάλτα, στην Κύπρο, την Ισπανία. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Διότι η Ιρλανδία, για παράδειγμα, δεν έχει να ανησυχήσει ε, από μεταναστευτικά κύματα προσφύγων, ούτε η Φιλανδία. Η Πορτογαλία ίσως τόσο. Θα πρέπει όμως, παρόλα αυτά, όλοι από κοινού να οργανώσουμε τον έλεγχο των συνόρων. Τώρα λοιπόν παραγγείλτε εσεί από το μενού αυτό. Τι θέλετε, τι θέλετε ακριβώ. Η Ευρώπη είναι το μόνο ε, επίπεδο που ουσιαστικά ε, δεν έχει χρέη. Υπάρχει απαγόρευση, απαγόλε απαγόρευση χρέους. Δήμοι, κοινότητε, περιφέρειες, τα κράτη-μέλη μπορούν να χρεώνονται και το έκαναν. Αλλιγότερο, αλ... περισσότερο αλλά πολλά τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί για όλους. Αλλά η Ευρώπη ε, για εμάς ε, πρέπει να είναι απαλλαγμένη από χρέη. Η υπερχρέωση δεν είναι ο δρόμος που θέλουμε. Απ' την άλλη δεν έχουμε φορολογικές αρμοδιότητες στην Ευρώπη. Ούτε μπορούμε να εισπράττουμε φόρους άμεσα. Το θέμα είναι ταυτόχρονα να βρούμε και τα μέσα και τα έσοδα για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε τις πολιτικές μας. Και τώρα έχουμε δύο τρύπε για το πολιετές της επόμενης δεκαετίας και ε, στην πλευρά των εσόδων και στην πλευρά των εξόδων. Παραδείγματο χάρη για το Brexit. Ε, επειδή ήταν καθαρίσεις φορείς οι Βρετανοί θα έχουμε 12 με 13 δις απώλεια τρύπα και στις δαπάνες επειδή έχουμε την άμυνα, την ε, προστασία των συνόρων, τη μετανάστευση, την ε, έρευνα. Αυτά θέλουμε ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μπορέσουμε να τα χρηματοδοτήσουμε. Για το κενό του Brexit προτείνουμε το 5% να γίνει με εξοικονομήσεις μέσω ε, του υπάρχοντος προϋπολογισμού και 50% νοπό χρήμα που θα προέλθει από τις 27 χώρες της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το άλλο, ε, την άλλη τρύπα των δαπανών, που μιλάμε εδώ για συμφέροντα ε, των πολιτών, αυτά τα προγράμματα που θέλουμε πρέπει να χρηματοδοτούν. Και λέμε 80% fresh money, νοπό χρήμα και 20% εξοικονόμηση από την αρχιτεκτονική του υφιστάμενου προϋπολογισμού στο πλαίσιο των κρατών μελών ήταν αρκετά αμφιλεγόμενες και επίμαχες οι συζητήσεις. Πέρα από λίγο ήμουν σαν κράτος μέλος και ο υπουργό Γεωργίας μου είπε κάνω ό,τι θες αλλά μην κόψεις τίποτα από τη Γεωργία. Μετά ήρθαν οι περιφερειακές αρχές και μου είπαν οι περιφερειάρχες μην κόψεις τίποτα από τη συνοχή. καμία περικοπή για 100 περιφέρειες και πάνω. Πρέπει όμως να προετοιμαστείτε. Δεν μπορεί να μην υπάρξει κάποια ε, περικοπή. Γιατί αλλιώς θα έχουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα έχει λίγα στολίδια πάνω, λίγα δώρα κάτω. Ούτε μπορούμε να καλύψουμε το Brexit βέβαια μόνο παραδείγματος χάρη με περικοπές γιατί αυτό θα ήταν λάθος. Θέλω την πολιτική συνοχή, θέλω ε, την γεωργία να μην τις βλάψω. Ναι, θα υπάρξουν κάποιες λογικές περικοπές. Αλλά θα ήταν λάθος να τσεκουρώσουμε αυτές τις ε, πολιτικές. 5-10%. Είναι κάτι που μπορούμε να το υποστηρίξουμε. 20-30 όχι. και θέλω επίσης ε, να υπάρχουν ε, οι δυνατότητες ε, για τη χρήση και αξιοποίηση των προγραμμάτων συνοχής από όλες τις περιφέρειες και όλες τις χώρες της Ευρώπης. Θέλω επίσης δύο προγράμματα στο μέλλον να μην έχουν καμία περικοπή, αντίθετα να αυξηθεί ο προπολογισμό. Το Erasmus Plus είναι το ένα για τη νέα γενιά, για την νεολαία και το Horizon 2020, μάλλον μετά το 2020, για την καινοτομία και για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Προετοιμάζει δύο εκθέσεις για το ΠΔΠ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι εδώ και οι δύο συγητές. θέλουμε να έχουμε ως όροφη, παραδείγματος για το ένα κενό, το 1,3%. Λένε κάποια κράτη-μέλη, όχι πλειοψηφία, μία μειοψηφία κρατών μελών. Λέει 1%. David Cameron. Ουσιαστικά έτσι τα βλέπει τα πράγματα. Αν μείνουμε στο 1, αλλά οι άλλοι θέλουν 1,3. Ποιος κερδίζει, ο Πούτιν, ο Ερντογάν και ο Τραμπ. Γιατί η Ευρώπη ε, θα είναι σχεδόν ακυβέρνητη. Θα χάσουμε τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Και έχουμε σημαντικά καθήκοντα, τα οποία δεν θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Εξού και παράκλησή μου προς όλους. Ας παραμείνουμε ευέλικτοι. Αν δεν είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς, ποτέ δεν πρόκειται να επιτύχουμε ομοφωνία στο Συμβούλιο. Εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί και να είμαστε όλοι έτοιμοι. Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Και Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν. Και ένα τελευταίο σημείο. Έχουμε την έκτη έκδοση. Ήταν ο Ζακ Ντελόρο πρώτος το 1988, το πρώτο πακέτο. αλλά το τι ίσχυσε επηρεάστηκε πάρα πολύ από τις ευρωεκλογέ που μεσολάβησαν. Ήταν τελείως διαφορετικό το πριν και το μετά. Δεν σημαίνει ότι μετά τα προβλήματα μπορεί να είναι λιγότερα. Μπορεί κανείς να λύσει κάποια προβλήματα χωρίς να κάνει τίποτα γιατί λύνονται από μόνα τους. Όμως αυτά τα οποία σας περιέγραψα εγώ δεν λύνονται από μόνα τους. Ούτε μπορούμε να φτάσουμε να συζητούμε το 2020 τι θα γίνει με τη Γεωργία, τι θα γίνει με τη διοίκηση, με την έρευνα, με τη Γεωργία. Θέλουν ξεκάθαρα πράγματα ήδη από τώρα. Και όσο το νωρίτερο τόσο καλύτερα. διότι Αντί να έχουν ολοκληρώσει το Μάρτιο 2011, χρειάστηκε για το προηγούμενο πλαίσιο οι συζητήσεις να πάνε μέχρι το 2013 και το 2014 ήταν μια χαμένη χρονιά. Αυτό δεν θέλουμε να συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος. Επομένως πρέπει να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας από τώρα μέχρι το Πάσχα του χρόνου Πρέπει λοιπόν αυτό το χρόνο τον να αξιοποιήσουμε για να συμφωνήσουμε μεταξύ μα και για να δώσουμε ξεκάθαρα μηνύματα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τις πολιτικές που ανέφερε. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Όλοι ακούμε, όλοι και περιμένουμε τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. Θα δώσω το λόγο στην Πρόεδρο κυρίως Γιάννοβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Πρέπει να εργαστούμε γρήγορα και Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών της ε, Βουλγαρίας, κυρία Μαρίνα Πετράνοβα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι ομιλώ εξ ονόματος της Βουλγαρικής Προεδρίας ε, ούσα αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών. Να εκφράσω τη στήριξή μας στον Επίτροπο Έτιγκερ και την απόλυτη συμφωνία μας μαζί του. Έχουμε συνεργαστεί με την Ουγγρική και την Αυστριακή Προεδρία για να εκπληρώσουμε από κοινού τον φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από το επόμενο Πάσχα. Πιστεύουμε ότι αυτή η προθεσμία είναι εφικτή είναι αυστηρή προθεσμία, σφιχτή, αλλά θα πρέπει όλοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Τούτων λεχθέντων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύθηκε στις 2 Μαΐου. Εμείς είμαστε, δημοσιεύεται στις 2 Μαΐου. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αμέσως με την επεξηγηματική φάση των διαπραγματεύσεων και να έχουμε σύντομες ή πιο ε, ε, ε, εκτεταμένες παρουσιάσεις στις μόνιμες αντιπροσωπεία αντιπροσωπείας των κρατών μελών στις Βρυξέλλες. Η πρώτη παρουσίαση μετά θα σχεδιάζουμε να γίνει στο Κορεπέρ και μετά τη δουλειά θα πάρει στα χέρια της ομάδα φίλων της Προεδρίας έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες συναντήσεις, όσο πιο ρεαλιστικό είναι αυτό, όσο το δυνατόν περισσότερες συναντήσεις ε, μπορούν να γίνουν, να γίνουν. Δηλαδή όχι παραπάνω από δύο συναντήσεις ε, το μήνα, για να μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε, να αρρωστικοποιήσουμε την φάση την επεξηγηματική και να περάσουμε πλέον με την Αυστριακή Προεδρία στην δεύτερη φάση. Και η πρόσφατη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες είναι πολύ υποστηρικτική. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε τη συζήτηση με αυτή την ανακοίνωση, να ε, τονίσουμε τις βασικές ε, οψιών, τις βασικές επιλογές, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να διαλέξουν την επιλογή που τους ταιριάζει καλύτερα. Άρα, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια ελαφρά αύξηση στις οροφές του πολιετούς δημοσιονομικού πλασίου γιατί έχουμε πολλές νέες πολιτικές που περιμένουν στην ουρά και πρέπει να εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις αλλά και οι μελλοντικέ, όπως είναι η μετανάστευση, η εξωτερική ασφάλεια, ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα και του καθεξής. Εν τω μεταξύ, θέλουμε και σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ των τριών, τριών βασικών λειτουργιών των δημοσίων οικονομικών. Δηλαδή, λειτουργία διανεμητική, λειτουργία χορηγητική και λειτουργία σταθεροποιητική. Ε, και θέλουμε να συμβάλλουμε και στις παραδοσιακές πολιτικές ε, ε, ενίσχυσης της συνοχής και του καθεξής. Όλα αυτά θέλουμε να αποκτήσουν την μέγιστη δυνατή σημασία και ε, για να τα επιτύχουμε πρέπει βεβαίως να συμπεριλάβουμε και τις νέες πολιτικές έτσι όπως παρουσιάζονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά έχω να πω προς το παρόν έτσι εν συντομία. Να σας πω ότι στο σήμα της Προεδρίας μας βασική προτεραιότητα είναι η συνοχή, μία από τις τρεις βασικές και φαίνεται αυτό και θέλουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά έτσι ώστε η πολιτική συνοχή να παραμείνει μία από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία από τις βασικές λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Πέτροβα. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Όλμπριχτ και στην κυρία Τομά. Συνεισηγητές για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο καθένας θα έχει 5-6 λεπτά στη διάθεσή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε οι συνεισηγητέ για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ ανήκω στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και η συνεισηγήτρια ανήκει στο στη Σοσιαλιστική Πολιτική Ομάδα και πάντοτε υποχρεωνόμαστε να βρίσκουμε ένα πολιτικό συμβιβασμό όχι μόνο μεταξύ ημών των δύο αλλά και με, με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα να εξηγήσω τη θέση μας. Ως Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν περιμένουμε να έρθει η σειρά μας στη διαδικασία. Αντιθέτως αντιδρούμε εξ αρχής και στο πρώτο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο δεύτερο και αυτή την εβδομάδα θα ψηφίσουμε την πολιτική μας θέση, την, τη θέση μας στην Επιτροπή για τον Προπολογισμό, την Κοινοβουλευτική και στη συνέχεια στην Ολομέλεια το ίδιο. Οπομένως αν η Επιτροπή έχει πρόβλημα με 27 υπουργού να ξέρει ότι θα έχει μεγαλύτερο με τους 700 τόσους βουλευτές μέλη από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ε, ε, γιατί δεν περιμένουμε τη σειρά μας τις εξελίξεις, αντιθέτως δρούμε εκ των προτέρων. Δύο είναι οι βασικές στρατηγικές. Είτε λέμε ότι, ε, είτε λέμε τι θα θέλαμε να κάνουμε και πόσο θα στοιχήσει αυτό που θέλουμε να κάνουμε και πού βρίσκονται τα χρήματα και ξεκινάμε με το τι θα θέλουμε να κάνουμε ή ακολουθούμε μία άλλη στρατηγική και λέμε ότι έχουμε τόσο τις εκατό και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το τόσο τις εκατό που έχουμε. Αυτές οι δύο στρατηγικές είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Η πραγματικότητα έχει ως εξής. Οι εθνικές κυβερνήσεις λένε ας κανονίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά λέμε θα δώσουμε χ τη 100 μόνο, 1%. Αυτό είναι αντιφατικό μεταξύ προτεραιοτήτων και οικονομίας, ενώ εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε διαφορετική θέση. Ερχόμαστε από πολλές διαφορετικές πολιτικές ομάδες και λέμε, οκ, αφού έχουμε τις προτεραιότητες έχει καλώς, αλλά υπάρχουν τα χρήματα για αυτές. Εάν όχι, πρέπει να ξανασκεφτούμε τις προτεραιότητες ή αλλιώ να δοθούν περισσότερα χρήματα. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε έχουμε πολιτικές ομάδες υπέρ της Ευρώπης που θέλουν να προσθεθούν περισσότερα χρήματα και υπάρχουν πολιτικές ομάδες ευρωσκεπτικίστριες που ή και κατά της Ευρώπης ξεκάθαρα που λένε αφού δεν υπάρχουν ε, χρήματα αρκετά ας κόψουμε προτεραιότητες και ας κόψουμε και μέρος του προϋπολογισμού. Άρα είναι σκληρή η συζήτηση, είναι δύσκολη η συζήτηση και τίθεται αυτό το ερώτημα. Τι θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο, ως Κοινοβούλιο θα προτείνουμε μια πολύ ρεαλιστική συμπεριφορά Δηλαδή, έχουμε ε, τα συγκεκριμένα πρότυπα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, ας μειώσουμε τον προϋπολογισμό με την συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου και ας μειώσουμε αυτό που παίρνει το Ηνωμένο Βασίλειο έτσι ώστε να αντισταθμιστεί η κατάσταση και να εξισορροπηθεί. Ωραία, αυτό το παίρνουμε ως σημείο εκκίνησης και λέμε από εκεί και πέρα τα της συνοχής να παραμείνουν ίδια, τα της γεωργίας να παραμείνουν ίδια, καμία μείωση εκεί στη συνοχή και στη γεωργία. Όμως ας τριπλασιάσουμε π.χ. το πρόγραμμα Erasmus Plus γιατί είναι πολύ σημαντικό και πολύ επιτυχημένο. Ας διπλασιάσουμε το COSME και το VA για τους νέους και τους ανέργους. Ας υπερασπιστούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και τη μετανάστευση. Και Ας ξεκινήσουμε από τη βάση της πυραμίδας πηγαίνοντα προς τα πάνω. Το αποτέλεσμα είναι 1,1 στα 3. Το 1,3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος είναι το προϊόν της δικής μας ανάλυσης. Και άρα εμείς τώρα ως Κοινοβούλιο θα πούμε στο Συμβούλιο «Καλώς, άμα δεν συμφωνείτε με αυτά που λέμε εμείς, ε, τότε εσείς τι προτείνετε να περικοπεί, τι θέλετε να αφαιρεθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δηλαδή από τι θέλετε να παρετηθείτε ως χώρες». Θέλετε να παρατηθείτε για παράδειγμα από τα, τους ελέγχους στα σύνορα. Θέλετε να παρατηθείτε από τα της έρευνας, από την συνοχή, από τη γεωργία και ποια θα είναι η αντίδραση του λαού σας τόπου, των πολιτών σας. Άρα ε, συνοψίζω και δίνω αμέσως το λόγο στη συνάδελφο Ιζαμπέλ Τομά και λέω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει τις πολιτικές ομάδες που και εσείς έχετε στα εθνικά κοινοβούλια, γιατί στα ίδια κόμματα ανήκουμε σε εθνικό επίπεδο. Ε, προσπαθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπροσωπήσει τις ίδιες πολιτικές οικογένειες και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ως εκπρόσωποι διαφορετικών πολιτικών οικογενειών λέμε στις κυβερνήσεις κυβερνήσεις να είστε ξεκάθαρε, πολύ σαφείς όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους Ευρωπαίους πολίτες να είστε σαφείς και σε αυτούς να πείτε στον κόσμο τι μπορεί να περιμένει γιατί αν ενισχύουμε συνεχώς τις προσδοκίες των λαών και τελικά δεν είμαστε αποτελεσματικοί, ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί. Παρόλο που έχουμε διαφορές μεταξύ μας σε αυτή την αίθουσα, το βασικό είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε την κοινή μας θέση και, να, ε, και λέμε ας είμαστε έντιμοι και ειλικρινεί για το τι πραγματικά περιμένουμε και θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ιζαμπέλ Τομά, συνεισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά. Για την Ευρώπη, όπως τελικά είναι κάτι που συμβαίνει και στην πραγματική ζωή, Καλές είναι οι δηλώσεις αγάπης και οι εκφράσεις αγάπης, αλλά κρατούν λίγο, δεν έχουν βάθος χρόνου. Το σημαντικό είναι τα διαπιστευτήρια, οι αποδείξεις αγάπης και η απόδειξη της αγάπης είναι τα λεφτά, ο προϋπολογισμός. Σήμερα πολλοί λένε και πολλοί εκδηλώνουν την αγάπη τους για την Ευρώπη, αλλά δεν δίνουν και πάρα πολλές αποδείξεις απτές για το πόσο την αγαπούν. Αυτά τα χρόνια πάρα πολλές φορές είχαμε περικοπές προϋπολογισμού. Το πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο είναι ε, χαμηλότερο από το προηγούμενο γιατί περιλαμβάνει την Κροατία χωρίς αυξήσεις. Στη συνέχεια είχαμε περικοπές ε, με τον πληθωρισμό. Κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός λόγω του πληθωρισμού είναι μικρότερος. Και παρόλα αυτά κάθε μήνα έχουμε τεράστιες διακηρύξεις, δηλώσεις, φιλοδοξίες, εκφράσεις για τη δημιουργία, για την ανάληψη νέων πρωτοβουλειών και νέων οραμάτων. Μα ζητούν να κάνουμε περισσότερα για τα σύνορα, για τις επενδύσεις, για την έρευνα, για το ένα, για το άλλο, αλλά με λιγότερα μέσα. Δεν είναι αυτό λογικό, ούτε δυνατό να γίνει. Κύριε Επίτροπε, ξέρω και πολύ καλά ε, το γιατί πράγμα μιλώ, γιατί έχω ηγητή από άλλη πολιτική ομάδα ομάδα. Επομένω, από, για, από συμβιβασμού ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Επίτροπε. Για να μπορεί να υπάρχει συμβιβασμό λοιπόν αποδεκτό από όλου, πρέπει όλοι να ε, λειτουργήσουν σωστά. Είναι προ το συμφέρον των κρατών μελών να δεχθούν, να διατηρήσουν τουλάχιστον τον προπολογισμό στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και όταν λέω να τον διατηρήσουν, με την αναχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα φτάσουμε όπως είπε και ο κύριος Όλμπριτς, είναι εισηγητής σε αυτό το 1,3% με την απλή διατήρηση των παραδοσιακών πολιτικών με ενίσχυση κάποιων βασικών εμβληματικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι το Εράσμος, η έρευνα και ορισμένες άλλες πολιτικές και με τις νέες πολιτικές. Και μόνο με αυτό ε, ε, φτάνουμε στο 1,3%. Με αυτά. Επομένως, θα ήθελα στη συνέχεια να μιλήσω για τη συνέχιση των κοινών μας δράσεων. Η κυρία Μαρινέλα Πέτροβα, η αναπληρώτρια υπουργό τη Βουλγαρική Προεδρία, μα είπε ότι θα έχουμε δύο συνεδριάσει το μήνα μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν. Χαιρόμαστε και σα συγχαίρουμε. Για την τακτή αυτή συνεργασία μεταξύ Κομισιόν και Συμβουλίου. Ωστόσο, τι έχετε προβλέψει για τις συζητήσεις με εμάς, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η διαδικασία είναι σαφής. Οφείλουμε στο τέλος της διαδικασίας να εγκρίνουμε και να συμφωνήσουμε με την πρόταση του Συμβουλίου την οποία θα έχει εκπονήσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκατάθεση σημαίνει συμφωνία. Συμφωνία σημαίνει συμβιβασμό. Συμβιβασμό σημαίνει συζήτηση. Πώς μπορούμε να δουλέψουμε μαζί και με τα εθνικά κοινοβούλια με τα οποία προσπαθούμε να συναντιόμαστε όσο τον ε, συχνότερα. Άρα τι έχετε προβλέψει για όλα αυτά. Και τέλος να είμαι και εγώ ε, πολύ ρεαλίστρια όπως είπε και ο κύριος Όλμπρεχτ και να πω το εξής. Κανείς δεν έχει το μαγικό ραβδάκι. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο να το διατηρήσουμε έτσι να μην το πάμε παραπάνω δεν μπορούμε συνεχώς να σκάβουμε και να αντλούμε πόρους από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Δεν είναι καλό πράγμα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς που έχουν δικές τους προτεραιότητες και δεν είναι καλό και για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνεχώς μειώνεται όπως είπα και προηγουμένως. Άρα πρέπει να επανέλθουμε στο πνεύμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, στην νοοτροπία του, δηλαδή να ξανασυμφιλειωθούμε με τους ίδιους πόρους. Και γι' αυτό αυτό το Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει και θα ψηφίσει υπέρ της δημιουργίας σύνδεσης μεταξύ του επομένου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου από τη μία και μιας πρότασης για τους ίδιους πόρους από την άλλη. Μιας πρότασης στην οποία έχουμε καταλήξει μαζί με τους αρμόδιους συνεισηγητές για τους ιδίους πόρους ακολουθούν μια ατζέντα ε, ταυτόχρονη και παράλληλη θα την ακολουθήσουμε μέχρι τέλους, μέχρι να δώσει το Κοινοβούλιο το πράσινο φως για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο ελπίζω κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ ότι το Συμβούλιο θα αλλάξει την ημερησία του διάταξη. Δεν είναι σοβαρό όταν νομίζει ε, ότι μπορεί να ε, έχει τη συνένεση ενός κοινοβουλίου που μόλις τώρα έχει εκλεγεί για παράδειγμα ενώ απέναντί του έχει μια κομισιόν η οποία έχει εδρεωθεί και έχει οριστεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να αλλάξει αυτή η μερίσια διάταξη, αυτός ο προγραμματισμός για να μπορέσουν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις το συντομότερο ε, δυνατό. Το χρονοδιάγραμμα δηλαδή πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Αρτουή, έχετε το λόγο για να διευθύνετε την ε, συνέχεια της συζήτησης. Ευχαριστώ κυρία Συμπρόεδρε. Ο λόγος στον κύριο Μαΐρ Αλκαγιά ε, που ε, συμμετέχει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Κατοχωρών. για πέντε λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας και όλους τους προσκεκλημένους και τους ομιλητές που μας παρουσίασαν την προοπτική τους για το, για το μέλλον του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Ήθελα να φωτίσω με διαφορετικό τρόπο ε, το όλο θέμα από την πλευρά του Ολλανδικού Σοσιαλιστικού κόμματο. Θέλω να δώσω έμφαση στα εξή δύο. Το πρώτο και πλέον σημαντικό είναι ότι ένα ευρώ στο πλαίσιο πρέπει να στηριχθεί από όλες τις κοινότητες όλων των κρατών μελών. Να είμαι ειλικρινή, κυρίε και κύριοι. Δεν είναι δεδομένο αυτό στι κατοχώρε. Μακάρι να μπορούσα να σας πω σήμερα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και συζήτηση ε, για την αποτελεσματικότητα και την ε, λογική των δαπανών του ευρωπαϊκού προπολογισμού, αλλά δυστυχώ υπάρχει. Και βεβαίω ε, και εγώ, σοσιαλιστή και ανθρωπιστή, δίνω μεγάλη αξία στην αλληλεγγύη. Όμω, αν δούμε ε, τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, το Ταμείο Συνοχή, τι κοινέ ευρωπαϊκέ πολιτικέ, ο κόσμο μα έχει αμφιβολίε. Αναρωτιέται αν η αλληλεγγύη και η αναδιανομή του πλούτου μπορεί να διοργανωθεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Το να αυξηθεί η συνεισφορά των ευρωπαϊκών χωρών προ τον ευρωπαϊκό προπολογισμό χωρί να αντιμετωπιστεί ο σκεπτικισμό των επιμέρου κοινωνιών και κοινοτήτων θα, θα ωφελήσει μάλλον μόνο του εθνικιστέ και όσου είναι κατά τη ε, διακρατική συνεργασία. Και ήδη βλέπουμε να αναδύεται κάτι τέτοιο και όχι μόνο στι κάτω χώρε. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη παρατηρήση μου. Το Brexit είναι μια μεγάλη ευκαιρία ε, υπό αυτή την άποψη. Έχουμε πολλές επιλογές ως ε, μέλος που, ε, όταν ένα κράτος μέλος που ήταν από τα ε, βασικά και από τους βασικούς συνεισφέροντες στον ευρωπαϊκό προπολογισμό να φεύγει. Δεν έχουμε μια προδιαγεγραμμένη τροχιά. Μετά από κάθε κρίση βλέπουμε να υπάρχουν όλο ένα και μεγαλύτερες ανάγκες για πολλούς η μόνη λύση είναι να ξεφύγουν από την ε, τροχιά αυτή και όχι να αφήσουμε το τρένο ανεξέλεγκτο, να, ακυβέρνητο, να συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα για το μέλλον της Ευρώπης και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να σκεφτούμε ότι ίσως να είναι καλύτερη μια μικρή Ευρωπαϊκή Ένωση όπου μερικά μόνο προγράμματα προτεραιότητας θα ε, λειτουργήσουν και ήδη η συγχρηματοδότηση μαζί με τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να είναι ο κανόνα και όχι η εξαίρεση. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα έπρεπε να περιοριστούν στο ελάχιστο. Ο προπολογισμό για ένα τέτοιο φιλόδοξο εγχείρημα, για αυτέ τι συγκεκριμένε φιλοδοξίε, θα έπρεπε να προσαρμοστεί αναλόγω μετά τον Brexit. Μόνο τότε θα είμαστε βέβαιοι ότι θα υπήρχε επαρκή στήριξη για ένα δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μα. Ε, περιμένω ε, τη συζήτηση που θα ακολουθήσει και σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Αλκαλιά. Και τώρα ο λόγος σε όσους από εσάς τον ζήτησαν. Δέκα έχετε ζητήσει το λόγο. Εάν μπορείτε να περιοριστείτε στο δίλεπτο, θα σας ήμουν ε, ε, βαθιά ευγνώμων. Πρώτος, ο κύριος Αντρέης Σλάτστα από την Πολωνική Βουλή. ίσως να είναι, να απόν αυτή τη στιγμή. Όχι, εδώ είναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός. Η πολωνική κυβέρνηση και το πολωνικό κοινοβούλιο παρακολουθούν τις όλες συζητήσεις για τον προπολογισμό και θέλουμε να τονίσουμε ότι σημαντικό είναι να δούμε τι έχει ήδη πετύχει στα πλαίσια της κοινή αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Θεωρούμε ότι όπως μόλις είπε ο Επίτροπος Έτιγκερ, η προστιθέμενη αξία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι υψηλή. Η πολιτική συνοχής έχει καλά δοκιμασμένα εργαλεία. Είναι λοιπόν άριστο μέσο για να πετύχουμε σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών. Θεωρούμε ότι αυτή η ψηλή προσταθέμενη αξία έχει να κάνει με τα έργα υποδομών. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση προς εμάς. Όταν συζητήσετε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, να θυμάστε να στηρίξετε με ευρωπαϊκά κονδύλια τέτοια μεγάλα προγράμματα όπως η Δία Μπάλτικα ή η Βία Κροάτσια. Να μην ξεχνάμε ότι είναι μεγάλα έργα αυτά υποδομών που αφορούν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολωνική κυβέρνηση και το πολωνικό κοινοβούλιο είναι πεπισμένοι ότι ό,τι προαθεί, προταθεί εντός της πολιτικής συνοχής μπορεί να προσφέρει. Μπορεί να είναι μια καλή απάντηση σε μεγάλες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως οι κλιματικές αλλαγές, οι, οι αλλαγές με την ε, κυκλική οικονομία, η τόνωση της ε, κοινοτομίας, η ψηφιακή αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος του Γιάνν Κράινερ από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Yes, uh, thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για να είμαι σύντομος. Θέλω να σχολιάσω μόνο το θέμα των ιδίων πόρων Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί φόροι και θα ήταν καλό τα κράτη-μέλη να δουν τι μπορεί να γίνει. Έχουμε το φόρο της κυροζήνης, για παράδειγμα, αν τον εφαρμόσει μόνο ένα κράτος, αυτό θα πλήξει την οικονομία του, το ίδιο για τον φόρο, με τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή το ενδεχόμενο επιβολής φόρου σε εκπομπές του άνθρακα, που θα έπλητε τις εθνικές βιομηχανίε, τα κράτη-μέλη, εάν δεν υπάρχει μια εναρμονισμένη προσέγγιση. Όταν λοιπόν το ευρωπαϊκό επίπεδο σκεφτείτε τους ίδιους πόρους θα πρέπει να σκεφτεί ε, ποιοι είναι οι, που θα, φόροι που θα μπορούσαν αυτοί να συλλεγούν από τα κράτη-μέλη αποτελεσματικά για να έχουν θετική επίπτωση κοινωνίες και στους πολίτες. Και έτσι θα αποκτούσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση τον απαραίτητο προπολογισμό για τα σημαντικά αυτά προγράμματα. Ιδίω εάν τα κράτη-μέλη δεν μπορούν ή δεν θέλουν να δώσουν τα χρήματα τα κράτη-μέλη. Ο Γενικό Εισηγητή ε, για τον Παγκόσμιο 2018, Ζίκφριτ Μούρεσαν, έχει τώρα το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, την κύριε αγαπητή συνάδελφη, είναι προφανές ότι πρέπει να ε, πρικοδοτήσουμε την Ένωση με ένα νέο πολιτές πλαίσιο που θα καθορίζει τη σχέση ε, μεταξύ πολιτών ε, και θεσμικών οργάνων της Ένωσης για την επόμενη δεκαετία. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν την ισορροπία μεταξύ παραδοσιακών προτεραιοτήτων, γεωργική πολιτική για παράδειγμα και πολιτική συνοχή. βοηθάει τις, πιο, ε, τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, ασφάλεια τροφίμων Έχουμε όμως και νέες προτεραιότητες ε, που παρέχουν περισσότερη ασφάλεια στους πολίτες, προστασία, να κάνουμε περισσότερα στην άμυνα και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την αντιμετώπιση της ε, προσφυγικής κρίσης, επένδυση στην ε, καινοτομία, να κάνουμε πιο ανταγωνιστική την Ευρώπη, προσανατολισμένη προς το μέλλον. Όλα αυτά πρέπει να τα εξορροπήσουμε μεταξύ τους. Χρειάζεται επίσης μεγαλύτερη ευελιξία. Το είδαμε αυτό όταν διαπραγματευόμασταν τον προπολογισμό του 2018. Είδαμε δηλαδή ότι το ΠΔΠ ε, αποφασίστηκε το 2013 για το 14-20. Τότε δεν ξέραμε ότι θα προκύψει η προσφυγική και η μεταναστευτική κρίση, ούτε οι τρομοκρατικές προκλήσεις ή οι απειλές για την ασφάλεια. Άρα τώρα πρέπει να προβλέψουμε πόρους για αυτά τα σημαντικά, που εξακολουθούν να είναι σημαντικά. Αλλά έχουμε να προσθέσουμε το ένα δις για τη συμφωνία με την Τουρκία, τα μέτρα για τη μετανάστευση, το ΕΦΣΙ, 200 δις επενδύσεων για τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Αντίστοιχο για την Αφρική. Άρα το βασικό μου μήνυμα είναι ευελιξία. Αλλιώ το 2024-2025 θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να πούμε στου πολίτε, αν προκύψει κάτι που δεν το είχαμε προβλέψει, ότι κινδυνεύουν αρχικέ μα προτεραιότητε. Και για να ολοκληρώσω, ακούω συναδέλφου, κύριε Πρόεδρε, που εκφράζουν ανησυχίε για το κατά πόσο θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο οι χώρες τους ε, στον ενωσιακό πλουσμό. Πρέπει όμως να γεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας. Τι θέλουμε να κάνει η Ένωση. Θέλουμε να κάνει πιο πολλά για την ασφάλεια, για τα εξωτερικά σύνορα, για την άμυνα, για την αντιμετώπιση τρομοκρατίας και το καθεξής. Εάν ναι, τότε πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα με πολύ λιγότερα. Φυσικά είναι σημαντική και η εφαρμογή φυσικά και χρειάζεται καλύτερη, ε, να, να κάνουμε καλύτερες ε, δαπάνες, πιο ορθολογικές. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα με πολύ λιγότερα. Άκουσα και τον προέρχεται από την Αυστρία. Αυτοί που δεν θέλουν να πληρώσουν ένα σέντ, η πραγματικότητα για αυτού είναι εξή. Αν θέλουμε να κάνει περισσότερη Ευρώπη, θα πρέπει να αυξηθεί με ένα μέτριο παθεί ορθολογικό τρόπο ο προπολογισμό. Ναι, πρέπει να πληρώσετε λίγο παραπάνω. Αλλά θα πάρετε και παραπάνω. Θα πάρετε αυτά τα ωφέλη κι εσείς και οι πολίτες σας. Αυτό που περιμένουν οι πολίτες από την Ευρώπη. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τα καθαρά ωφέλη, δεν θα είναι χειρότερα τα κράτη-μέλη παρά το ότι κάποιοι αυτό νομίζουν. Ευχαριστώ. Merci. La parole est maintenant à... Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Ματίας Βίρτ που είναι από την Οικρική Βουλή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους βουλευτές. Έχουμε μπροστά μας μια σειρά από νέες προκλήσεις και ιδίως το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με 12-13 δις ευρώ λιγότερο που θα προκύψουν από το Brexit. Έχουμε όμως να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερες προκλήσεις στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και την προβλεπόμενη διεύρυνση με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν θέλουμε να πλήξουμε την κοινή αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχή. Πρέπει να υπάρξουν ε, πιο γενναίες συνεισφορές από τα κράτη-μέλη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις πολιτικές μας για να υποστηριχθεί η συνοχή μας και η ανταγωνιστικότητά μας. Είναι ε, προτεραιότητες αυτές και ε, τα ωφέλη θα είναι σημαντικά για τις χώρες που συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία επικοινωνία επιτρέπει να καλύψουν τη διαφορά οι χώρες που είναι πιο μακριά από τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Άρα, μακροπρόθεσμα, μπορεί να μειωθούν τελικά οι φορές Γι' αυτό πρέπει πρώτα να ορίσουμε σαφείς προτεραιότητες και μετά να προσαρμόσουμε αναλόγως τους δημοσιονομικού μας, δημοσιονομικούς μας πόρους. Πρέπει να προετοιμάσουμε ένα πλαίσιο που να είναι εύληπτο, διαφανές και εποφελές για όλους. Η Ουγγαρία είναι πανέτοιμη είναι πανέτοιμη να συζητήσει τη συνεισφορά της για την περίοδο μετά το 2020. Ίσως να πάμε και παραπάνω από το 1,1 του ΕΠ. Γι' αυτό όμω χρειάζονται προτάσεις ε, πολύ καλά επεξεργασμένες και σαφείς. Δεν θέλουμε καθυστερήσεις στην έγκριση του πολίτης δημοσιονομικού πλαισίου. Θα ήταν θετικό, καλό να προβλεφθούν συγκεκριμένε καταληκτικέ ημερομηνίε, ώστε και το Ευρωκοινοβούλιο να μπορεί να κάνει τη δουλειά του ε, ως συνομοθέτης όπως πρέπει. Για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ε, νομική βεβαιότητα, βεβαιότητα δικαίου και ως προς την σωστή κατανομή των πόρων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Ηλίας Μυριάντος από την Κυπριακή Βουλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομολογουμένως ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχουν λεχθεί από τον Επίτροπο κύριο Νέτιγκερ και παράλληλα θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων στη διαμόρφωση του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για απολετελεσματικότερη αντιμετώπιση των κρίσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής βοήθειας προς τα πληγέντα κράτη μέσω των προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πολύ εύστοχα έχει επισημαίνει ο κύριος Επίτροπος. Η αρχή της αλληλεγγύης πρέπει να ενσωματωθεί και να ενισχυθεί στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σχεδιασμών για τη διαμόρφωση της νέας κοινή γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής μέσα μετά το 2020, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πώ προστατεύονται αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα και πώ διασφαλίζονται τα ευρωπαϊκά ενεργειακά αποθέματα όπω αυτά έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα στην ε, κυπριακή αός και πώ αποτρέπονται κάποιε ε, χώρε να ενεργούν αντίθετα προ τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. παράλληλα όμω η ευρωπαϊκή ένωση μέσα από το ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να στηρίξει αποτελεσματικά επενδύσεις για την εκμετάλλευση των δικών της ενεργειακών αποθεμάτων. Παράλληλα, θα έλεγα ότι η κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχή διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόθεση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στη μείωση των ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Συνεπώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές αυτές παραμένουν ψηλά στις προτεραιότητες του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και ότι θα διατηρηθεί το μερίδιο του πλαισίου αυτού που επενδύεται σε αυτές. Ε, Επίση, συμφωνούμε με τις θέσεις της Βουλγαρικής Προεδρίας για τη διατήρηση αυτής της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Συνοχής. Στις επικείμενες επίσης συζητήσεις σχετικά με τον μηχανισμό κατανομής μελλοντικής πολιτικής ε, για τη συνοχή πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα κριτήρια που να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ε, ιδιαιτερότητες ιδιαίτερα όσον αφορά τις απομονωμένες νησιωτικές ε, περιοχές. και τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εγγύηση για την νεολαία και απασχόληση των νέων, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία νέων ποιοτικών αξιοπρεπών θέσεων, πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. Επίσης, τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και προγράμματα για την κατάρτιση που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να διασυνδέονται και με τις ανάγκες αγοράς και υπογραμμίζω τέλος την ανάγκη ρύθμισης κενών που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία, τη βελτίωση των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων, σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Συνεργασία και την κοινωνία των πολιτών και του κοινωνικού Εταίρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ο κ. Παπαδημούλης. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει, όπως είπαν και οι συγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον νεοπολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να επενδύσουμε περισσότερα και περισσότερο στο κοινό μας μέλλον και από αυτό θα κερδίσουν όλα τα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη που είναι καθαροί εισφορείς. Γιατί είναι αδύνατον να κάνουμε περισσότερα μαζί με λιγότερα χρήματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι και το ποσοστό του 1,3% είναι το ελάχιστο που πρέπει να συμφωνηθεί από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου και αυτή η αραγής ενότητα του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να μείνει μέχρι τέλους και νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε πολιτικές όπως το Erasmus Plus ή το Horizon, να μην μειωθεί ούτε ένα ευρώ το κονδύλι που προβλέπω για τις πολιτικές συνοχής και για την κοινή αγροτική πολιτική και επειδή έχουν προσθεθεί και καινούργιοι στόχοι για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, της τρομοκρατικής απειλής, πρέπει και τα κράτη-μέλη να δώσουν περισσότερα γιατί θα τα πάρουν στο πολλαπλάσιο από ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια και να υιοθετήσουμε δύο-τρεις τουλάχιστον καινούριου νέους πόρους με κοινέ ευρωπαϊκές πολιτικές. Φορολόγηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος ή της κυροζίνης ή του φόρου για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μπορεί να δώσουν σημαντικά έσοδα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και την ίδια ώρα να αποφύγουμε το φορολογικό ντάμπινγκ. Κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν κατευθείαν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι απλώς πρέπει να στηρίξει τις, τις προτάσεις της Κομισιόν, αλλά να είναι πιο φιλόδοξο και πιο απαιτητικό, έτσι ώστε να αντιρροπήσει τις πιέσεις ορισμένων κρατών μελών οι οποίες έχουν μια πολύ εγωιστική προσέγγιση απέναντι στην κοινή ευρωπαϊκή μας προσπάθεια. Θέλουν να δίνουν λίγα και να τα παίρνουν όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαστάη Κούρας από την Βουλή των Ελλήνων. Κύριε Πρόεδρε, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αντιμετωπίζει πολλές νέες προκλήσεις προκλήσεις που απαιτούν ένα νέο, διαφανή, απλό, ενισχυμένο και σύγχρονο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έγκαιρα όμως συμφωνημένο. Πλαίσιο αυξημένης λογοδοσίας, ευέλικτης διάρθρωσης, στοχευμένο σε τομείς αυξημένης προστιθέμενης αξίας και σημαντικής μόχλευσης. Τι να περιλαμβάνει όμως το μενού αυτού του πλαισίου όπως ρώτησε ο κ. Επίτροπος. Όπως σωστά ανέφερε η κυρία Πέτροβα, την επιτέλεση καταρχήν των βασικών λειτουργιών, όπως είναι οι επενδύσεις σε δημόσια αγαθά, η αναδιανομή και η μακροοικονομική σταθεροποίηση. Κίνητρα στα κράτη-μέλη για την υλοποίηση διαθεωτικών μεταρρυθμίσεων. Ενίσχυση της αλληλεγγύης, της δημιουργικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και της αιρεσιμότητας μεταξύ χρηματοδότησης και σεβασμού θεμελιωδών αξιών, όπως είναι το κράτος δικαίου ενίσχυση των πόρων για τη μετανάστευση και το άσυλο, ειδικά σε μια περίοδο άνισα κατανεμημένων μεταξύ των κρατών μελών μεταναστευτικών ροών. Αμετάβλητους πόρους για την κοινή αγροτική πολιτική και την πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη. Επαρκείς πιστώσεις σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, σε δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας, σε τομείς όπως είναι η προστασία των εξωτερικών συνόρων, η ενίσχυση της νησιωτικότητας, η στήριξη της κινητικότητας των νέων και η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Και τέλος, προφανώς γιατί πρέπει να δούμε και το θέμα των εσόδων, η αξιολόγηση του υφιστάμενου τρόπου χρηματοδότησης του πλαισίου με την προσθήκη νέων πόρων που θα δώσουν βιώσιμη λύση στο ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Νταν Μπάρτνα τώρα, από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα η συζήτηση που έχουμε φυσικά και αφορά ε, την ε, κατάρτιση του περιπολισμού για το μέλλον, αλλά είναι και μια βαθύτερη συζήτηση για το μέλλον των οικονομικών της Ευρώπης. Μια πρώτη ιδέα είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια επανειεράρχηση των πολιτικών ε, προτεραιοτήτων σε συνάρτηση με τον περιβολισμό, χωρίς αυτό όμως να αυξήσει το χάσμα μεταξύ καθαρών εισφορέων και καθαρών δικαιούχων. Πρέπει να μειώσουμε τις ανισότητες και όχι να εμβαθύνουμε αυτές και να μεγαλώσουμε το χάσμα. Επίσης πρέπει να υπάρχει και δημοκρατικός έλεγχος ε, των ε, οικονομικών. Οι πολίτες ε, δεν εμπιστεύονται τις οικονομικές, δημοσιονομικές πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη, να καταστήσουμε πιο σαφές αυτό το πολύπλοκο σύστημα. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Βέβαια, στο μέλλον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους. Το Brexit Φυσικά και σημαίνει μείωση του ενωσιακού προπολογισμού μετά το 20 ιδίω. Αυτή η τρύπα όμως θα πρέπει να κλείσει, αλλά κατά τρόπο που δεν θα ασκηθούν περισσότερες πιέσεις στα κράτη-μέλη. Πρέπει να βρεθούν νέοι ήδη πόροι. Ιδίως για τις πολιτικές νέας γενιάς, όπως είναι ψηφιακή οικονομία, έρευνα και ανάπτυξη. Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει απλούστευση των μηχανισμών στο προσεχές ΠΔΠ και να εντοπιστούν και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την προσέλκυση κεφαλαίων που θα βοηθήσουν τη διαφοροποίηση των ιδίων πόρων της Ένωσης για να μπορεί η Ένωση να αντιμετωπίσει περισσότερο τις αναδυόμενες προκλήσεις όπως είναι η μετανάστευση, η ασφάλεια στο πλαίσιο το επόμενο. Επίσης πρέπει να είμαστε πιο καινοτόμοι και ευέλικτοι, συμφωνώ. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι το προσεχές ε, πι θα καθορίσει κατά πάσα πιθανότητα και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί στο μέλλον η Ένωση ως καταφύγιο. Σίγουρα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητες στις πολιτικές νέας γενιάς της Ένωσης, όπως είναι η ψηφιακή οικονομία ή η ενιαία ψηφιακή αγορά, αλλά θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή και στις παραδοσιακές πολιτικές κάτι που θα ωφελήσει όλες τις χώρες, γιατί πάνω σε αυτές δράστηκε και εξακολουθεί να δράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τις ενισχύσουμε, να προσαρμόσουμε, όπως χάρη την πολιτική συνοχή και την ε, κοινή πολιτική στις νέες πραγματικότητες και να παραμείνουν στον ορίζοντα μετά το 2020 προτεραιότητα αυτές τις πολιτικές. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Σοφία Ριμπέιρο τώρα από το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βρίσκομαι εδώ στα δεξιά σας. Ο Επίτροπος Αιτιγκέρα έκανε μια έκκληση, απίθυνε μια έκκληση για μεγαλύτερη ευελιξία του Κοινοβουλίου και γενικώ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για την ε, διαπραγμάτευση που προβλέπεται για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή η έκκληση έχει να κάνει με τις απαιτήσει ασφάλειας και τους περιορισμούς που επιβάλλει το Brexit. Είναι σημαντικό αυτό και στην ανακοίνωση που μας ε, υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα για τους στόχους της και τα διάφορα σχέδια που προβλέπονται στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, στα κεφάλαια της πολιτικής συνοχής και της ΚΑΠ. Εκεί το σενάριο, το το οποίο που προβλέπετε, ότι δεν θα υπάρχει η ίδια χρηματοδότηση, ιδίω στην ΚΑΠ. Θέλετε να προβλέπετε ε, μείωση στη χρηματοδότηση μέχρι και 30%, κάτι που θα είναι πραγματικά καταστροφικό για ορισμένε περιοχέ. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι στόχοι τη ΚΑΠ είναι στόχοι που αυτή τη στιγμή επηρεάζονται από τους ήδη επιβεβλημένους περιορισμούς τις περικοπές που θα εντατικοποιηθούν. Ε, οι κειμενόμενες τιμές στην αγορά, ε, το θέμα της ε, τροφικής αλυσίδας, το θέμα των νέων προκλήσεων δημιουργίας αλυσίδων παραγωγής αξίας, της επιστηστικής επάρκειας των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξη, ακόμη και των στόχων προστασίας των τιμών για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές. Εάν δεν γίνει μια τεκμηριωμένη, εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων αυτών, ακόμη και στο γενικό πλαίσιο, και αφήσουμε την ΚΑΠ να είναι φτωχό συγγενής στον προπολογισμό της Ένωσης, να διατηρηθούν άλλε πολιτικέ τη Ένωση ει βάρη τη γεωργία δηλαδή, νομίζω ότι έτσι υποβαθμίζουμε γενικώ τι οικονομικέ συνθήκε, τι κοινωνικέ συνθήκε, διότι η χρηματοδότηση τη γεωργία ε, έχει απευθεία αντίκτυπο στο 90% τη ε, ευρωπαϊκή επικράτεια που είναι επικράτεια τη ε, υπαίθρου, είναι ύπεθρο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε συνάδελφε. Και τώρα ο κύριο Μπαλαούρας από την Ελληνική Βουλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέρσι στη Ρώμη οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έβαλαν στόχο για Ευρώπη πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική, με οικονομική και κοινωνική σύγκληση και συνοχή. Για να υπάρξουν όμως αυτές οι ευχές πρέπει να υπάρξει πολιτική θέληση. Μια βάση δηλαδή που μας δηλώνει ότι είναι η δημοσιονομική επάρκεια. Ο αρμόδιος επίτροπος όμως πρότεινε περικοπές δαπανών για την κοινή αγροτική πολιτική, για παράδειγμα μείον 5% και, για την πολιτική συνοχή σε διαθροτικών ταμείων μείον 10%. Η συζήτηση υπήρξε, αλλά μετά το Brexit εντάθηκε. Ποια είναι η λύση και άλλες μειώσεις στην ΚΑΠ κοινή αγροτική πολιτική και στα διαφροντικά ταμεία στο 20% όπως υπάρχουν εισηγήσει. Πότε, τώρα κύριε Πρόεδρε που είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο αυξημένων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, μειωμένων επενδύσεων και μεγάλης ανεργίας, κοινωνικού αποκλεισμού και αυξημένων μεταναστευτικών ορών. Προτείνουμε να μην να μην κοπεί χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχή να αυξηθεί η στήριξη στις λιγότερα αναπτυγμένες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα απομόνωσης νησιωνικότητα βιομηχανικής παρακμής. για το μεταναστευτικό υπάρχει πρόβλημα θα κλείσουμε ξανά τα μάτια και όσον αφορά το οικονομικό ζήτημα πρέπει να ενισχυθούν τα κράτη εκείνη που δέχονται τις ε, μεταναστευτικέ ροέ, αλλά ταυτόχρονα να υπάρξει και δίκαιη κατανομή. Τέλος, ερώτηση που γίνεται και από τους ε, συναδέρφους εδώ αλλά και από εσά είναι από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Εχθέ κάναμε μια ολόκληρη κουβέντα για την φοροαπηφυγή τεραστίων κολοσσών, μεγάλων κολοσσών έτσι που αποφεύγουν να πληρώνουν ε, φόρους για να φτιάξουμε ενιαία φορολογική πολιτική για να αποφύγουμε τελικά το κοινωνικό και οικονομικό ντάμπινγκ διαφόρων κρατών. Να συζητήσουμε μεταξύ μας οι χώρες για τη σημερινή διάθρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, προχτές βγήκαν στοιχεία ότι η Γερμανία έφτασε το πλεόνασμά της στο 8,1% ε, του ΑΕΠ. Εμείς κύριε Πρόεδρε χρειαζόμαστε ένα σύμφωνο για την απασχόληση την ανάπτυξη με νέες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές υπέρ των, του λαού, των λαών. Δημόσιες επενδύσεις που θα εισακτούν στην πραγματική οικονομία για να δώσουν δικαιώματα στους εργαζόμενους. Αναθεωρημένος ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης με κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα που θα ενισχύσουν την κοινωνική και οικονομική σύγκληση και συνοχή και τέλος, οι σημερινές πολιτικές που έχουν βλάψει πράγματα την Ευρώπη και έχουν συμβάλει στην άνοδο της ακροδεξιάς και των ξενοφοβικών δυνάμεων απειλούν τη δημοκρατία και την ειρήνη. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν την πορεία μας, να επιβάλλουμε κοινωνική και περιφερειακή σύγκληση και συνοχή για την αηφόρο, οικολογική και χωρίς αποκλεισμού Merci. ευχαριστούμε και τώρα ο Γιώργεν Άντερσον από τη Σουηδική Βουλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα εκπλαγείτε αν έχετε ήδη ακούσει ότι η γενική θέση της Σουηδίας είναι ότι θα θέλαμε πιο περιορισμένη δημοσιονομική πολιτική. Η σημερινή συζήτηση είναι κέρια καλώς συζητούμε τις απόψεις μας, το τι πιστεύουμε, ώστε να έχουμε κάποια εικόνα για το τι θέλουμε να προκύψει από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Υπάρχουν πολλά σημαντικά που πρέπει να χρηματοδοτήσουμε, να τα προσπαθήσουμε και να τα επιδιώξουμε από κοινού. Όμως το επίπεδο φιλοδοξιών που θέλουμε να πετύχουμε με τον προπολογισμό είναι πολύ διαφορετικό αν ακούσουμε τους διάφορους συναδέλφους εδώ στην αίθουσα. Νομίζω είναι καλά τα θέματα που συζητούνται, όμως υπάρχουν ε, θέματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με άλλο, από άλλη οδό. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι θέλουμε και χρειαζόμαστε την προσφορά ευημερία, στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωση μέσα από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ενώ άλλοι λένε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι 350 δις, αλλά με τις τάσεις που έχουν διαμορφωθεί βλέπουμε, πεντα... βλέπουμε τη δυνατότητα να έχουμε 500 δις παραγωγή κέρδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι υπερεκτιμώνται κάπως οι δυνατότητες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ως προς την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την ε, καλή απόδοση ευημερία. Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε από κοινό πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα την ενιαία αγορά, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον προστατευτισμό εντός της Ευρωζώνης. Νομίζω ότι θα είναι πιο σοβαρή η επίπτωση που θα έχει κάτι τέτοιο στο να ανακατανεμηθεί σωστά ο πλούτος. Θα ήταν και ενδιαφέρον για τις εταιρείε των πλουσιότερων χωρών να ε, μετατοπίσουν τις εταιρείε τους στις χώρες που είναι φτωχότερες. Είναι απλό και είναι ένας τρόπος να ανακατανεμηθεί έτσι ο πλούτος. Αυτό είναι ένα βήμα προόδου που μπορούμε να κάνουμε. Είναι ήδη καλό το ότι τα συζητάμε όλα αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε ο κύριος Ιβάνοφ από τη Βουλγαρική Βουλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, και τώρα περνάω στα βουλγαρικά. Η συζήτηση η οποία λαμβάνει χώρα όχι μόνο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και σε άλλα βήματα συζήτησης είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να συναγάγουμε το συμπέρασμα ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση για να είναι μεγαλύτερη η ισότητα μεταξύ τους. Επειδή μιλάμε για φόρους, έκανε μια έρευνα το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το αποτέλεσμα ήταν ότι λόγω της φοροδιαφυγής από το ΦΠΑ 150 δισεκατομμύρια ευρώ δεν μπαίνουν στα δημόσια ταμεία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το δούμε και αυτό. Πρέπει να δούμε τον τομέα του ΦΠΑ όταν μιλάμε για αύξηση των εθνικών εισφορών. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω, δυστυχώς δεν είναι πλέον παρόν ο Επίτροπος Έτιγκερ. Μίλησε για συμβιβασμό. Φυσικά και πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ όλων των κρατών μελών. Όμως, Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ότι ένα σύστημα είναι τόσο ισχυρό όσο ο πιο αδύναμος κρίκος του. Γι' αυτό λοιπόν ενθαρρύνω όλες και όλους να συνεχίσουμε με την πολιτική συνοχή και όλες τις πολιτικές που αναφέρθηκαν με την ίδια χρηματοδότηση, να μην μειωθούν τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τη συμμετοχή σας ε, στη συζήτηση αυτή. Και επειδή έχουμε ακόμη λίγο χρόνο, μέχρι τις 5 και 4 οπότε πρέπει να κλείσουμε, στρέφομαι στους συνεισηγητές μας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020, την κυρία Τόμα και τον κύριο Όλμπριχτ. Και το ζητώ να εφερολογήσουν αλλά σύντομα. Κυρία Τόμα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι θα είμαι πολύ σύντομη, διότι όπως και οι συναδελφοί μου από τα Εθνικά Κοινοβούλια, έτσι και εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή ήταν πάρα πολύ πλούσια, άκρος ενδιαφέρουσα και τα όσα άκουσα μου δημιουργούν την εντύπωση ότι δεν απέχουμε πολύ από το να είμαστε σε ένα βήμα συζήτησης ε, που έχει ε, εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, κάπου αλλού και θα πει θα, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε πολύ εύκολα μεταξύ μας. Αφού μπορούμε μεταξύ μας λοιπόν να συμφωνήσουμε γιατί να μην προσπαθήσουμε να πείσουμε καθένας τα μέλη της κυβέρνησής του. Εμείς θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή όσο χρειαστεί με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ. Συμφωνώ με την άποψη ότι η συζήτηση αυτή είναι κάπως διαφορετική σε σχέση με προηγούμενες ε, συζητήσεις που είχαμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αφού να πω ότι πολλές φορές είχαμε καθαρέθιμο τυπικές ε, συζητήσεις σίγουρα αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, για να μην πω κρίσεις, και είχαμε δύσκολες προκλήσεις ε, και δύσκολες επιλογές να κάνουμε. Βλέπουμε όμως ότι η διαφορά προσέγγισης δεν έχει να κάνει με τη διαφορά των πολιτικών ε, κομμάτων, αλλά με τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν κάποιοι που λένε το ίδιο ακριβώς με τις κυβερνήσεις τους και είναι πολύ σημαντικό να το σημειώσουμε αυτό. Δεύτερον, οι εθνικοί βουλευτές και εμείς εκλεγόμαστε από τους πολίτες, από το λαό και σε αυτούς είμαστε υπόλογοι και πρέπει να εισακουστούν οι επιθυμίες τους και αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς. Αν οι πολίτες μας φοβούνται και θέλουν ασφάλεια, αν αυτό για αυτούς είναι το πιο σημαντικό, πρέπει να είναι και για μας το πιο σημαντικό. Αν μας ρωτάει ο κόσμος, προστατεύετε τα σύνορα, θα πρέπει και εμεί να θέσουμε το εξή ερώτημα. Έχουμε επαρκεί πόρου για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα προστασία των συνόρων. Αν δεν το γνωρίζετε, δείτε το έγγραφο τη Κομισιόν τη προηγούμενη εβδομάδα. Θα διαβάσετε εκεί ότι η Κομισιόν λέει εξαρτάται από το τι θέλετε. Τα λέω από μνήμη βέβαια. Λέει, αν θέλουμε μια στενή προστασία των συνόρων, ωραία μπορούμε να έχουμε 5.000 στρατιώτες, αλλά αν θέλουμε να έχουμε καλύτερη προστασία θέλουμε 20.000 αν θέλουμε να το κάνουμε όπως οι Αμερικανοί, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 100.000. Τουλάχιστον 100.000. Ας είμαστε σοβαροί λοιπόν. Είτε θέλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορα, οπότε θα χρειαζόμαστε 80 ή 100.000 στρατιώτες, αλλά πού είναι τα χρήματα γι' αυτό. Οι ψηφοφόροι μας τι θέλουν, θέλουν να τους προστατεύσουμε. Αν θέλουν να τους προστατεύσουμε, με ποιο τρόπο θα το κάνουμε. Έχουμε τις παραδοσιακές πολιτικές, γεωργία, πολιτικές συνοχής. Στο μυαλό πολλών πολιτικών αυτό θα πει παράδοση. Για πάτε όμως στην Πολωνία, τη Βουλγαρία, Τσεχία. Θα δείτε εκεί ότι η πολιτική συνοχή πολύ συχνά αφορά την έρευνα, την καινοτομία. Δεν αφορά μόνο δρόμους, αφορά τη σύγκληση σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Δεν θα πει παραδοσιακή συνοχή ε, δημιουργώ πισίνες, ε, φτιάχνω πισίνες, γιατί βέβαια αυτό είναι κάτι που όλοι είναι αντίθετοι εφόσον πρόκειται για σπατάλη χρήματος. Αλλά μιλάμε για άλλου είδου επενδύσεις εδώ. Σε εφείς υποδομές για παράδειγμα και αυτό είναι διαφορετικό. Θέλω να σχολιάσω κάτι που είπε ο Σουηδός ε, συνάδελφος. Όλοι κάνουμε υπολογισμού και λέμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα με τον ενωσιακό προπολογισμό. Δεν είμαστε ειλικρινεί όμω με τον κόσμο. Πώς θα μειωθεί η νεανική ανεργία. Θα μειωθεί με αυτόν τον ε, προϋπολογισμό που έχουμε. Όχι, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ας ξεκινήσουμε κάποιες δραστηριότητες για να έχουμε αυτή ε, τη μόχλευση, για να δώσουμε κίνητρα, διευκόλυνση. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα με τη μια, γιατί αν το πούμε αυτό, συγγνώμη που το λέω, λέμε ψέματα. Ψευδόμαστε όταν λέμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Είναι λοιπόν τώρα η ώρα για όλους μας να είμαστε σοβαροί και να είμαστε συγκεκριμένοι. Γιατί ο κόσμος περιμένει από εμά να είμαστε ξεκάθαροι για το τι θέλουμε, για το τι μπορούμε να κάνουμε και για το τι είναι εφικτό να γίνει. Και όπως είπε και η Ζαμπέλ Τομά, εμείς το Κοινοβούλιο και εμείς οι δύο όσοι συγκητές είμαστε στη διάθεσή σας ε, και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί σας οτιδήποτε θεωρείτε ότι πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο αυτής της ε, διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Γιάνν Όλμπριχτ, ευχαριστούμε Ιζαμπέλ Τόμα, ευχαριστώ τον καθένα από εσά ξεχωριστά. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της... Α, θα τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διευθύντρια επί των Προπολογισμών. Κυρία Καβιό. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του Επιτρόπου Έτιγκερ, ο οποίος έπρεπε να φύγει γιατί είχε κάποια ανεκμένη υποχρέωση. Δεν πήρα το λόγο προηγουμένως, όμως νομίζω ότι χρήσιμο θα ήταν να ε, προσκαλείτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητά μαζί σας, να απαντά σε ερωτήσεις εφόσον έχετε και όπως είπε ο κ. Όλμπριχτ, μόλις την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσίευσε μια ανακοίνωση που θα συνεισφέρει στις συζητήσεις των αρχηγών κυβερνήσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή και σας ευχαριστώ όλους για τη μεγάλη σας ενδιαφέρον ε, για τα θέματα αυτά και από τις Εθνικές Βουλές και από το Ευρωκοινοβούλιο. Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε όποια ερώτηση έχετε για το έγγραφο αυτό και για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ κύριε Αρτουή που μου δώσατε την δυνατότητα να απαντήσω. Merci. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Καλβινιό. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας. Φτάνουμε στο τέλος αυτού του μέρους της συνάντησής μας. Πλούσια συζήτηση και είδαμε πόσο έχουμε κοινέ ευθύνε. τόσοι βουλευτές από τις Εθνικές Βουλές και εμεί ε, στο Ευρωκοινοβούλιο. Κοινέ ευθύνε και οικονομική υφή και δημοσιονομική. Η ευθύνη που μα έχει ανατεθεί να σχεδιάσουμε την επόμενη φάση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου μας ε, καλεί να λάβουμε αποφάσει για την περίοδο 2020-2027. Πραγματικά δυσκολεύομαι να σας δυσκολεύομαι να, να φανταστώ ότι θα συμβεί το 2025, ή 2027. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που τρέχει τώρα, 2014-2020, ε, πέρασε από πολύ δύσκολες ε, δοκιμασίες ε, όταν αντιμετωπίσαμε διάφορα φαινόμενα κρίσης, την μαζική μετανάστευση του 2015, όταν βρισκόμασταν στην φάση αδυναμίας στην Ευρώπη. Ήταν δύσκολο να φανταστούμε ότι θα δημιουργηθεί ένα ολόκληρο ε, γαλαξίας του προπολογισμού με τους διάφορους δορυφόρους που χρειάστηκε να προβλέψουμε θα πρέπει λοιπόν να πείσουμε τους πολίτες, να καταλάβουν μέσω του προπολογισμού ποιες είναι οι φιλοδοξίες μας, ποιο είναι το όραμά μας για το γίγνεσθε αυτής της Ευρώπης που θέλουμε από κοινού να οικοδομήσουμε, για να ε, οπλιστούμε για το μέλλον, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση στους κινδύνους που παρουσιάζει υπό κάποια έννοια. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε αυτή τη βαθιά ευθύνη και έχουμε και ένα επιπλέον ρόλο διότι ο προπολογισμό αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται από του ιδίου πόρου που κυρίως είναι τελωνιακοί δασμοί. Τελωνιακοί δασμοί που είναι 10% των ε, πόρων του προπολογισμού. πού έρχονται το 90% από τους εθνικούς προπολογισμού. Δηλαδή εσείς ψηφίζετε τους πόρους. Εμείς έχουμε ευθύνη μόνο για τις δαπάνες τις ε, δαπάνες όμως που είναι ικανές και αναγκαίες και που μπορούν να προσφέρουν κάτι. Καταλαβαίνετε πόσο αναγκαίοι είναι ήδη οι πόροι λοιπόν, αλλά αν ε, διαβάσουμε την έκθεση του κυρίου Μόντι που προείδευσε στην ομάδα ψηλοπιπέδου για τους ίδιους πόρους, οι πόροι, οι νέοι ίδιοι πόροι, δεν έχουν σκοπό να δημιουργήσουν και νέους πόρου προπολογισμού, κάτι το πρόσθετο. Ο σκοπό είναι να μειωθεί η συνεισφορά των κρατών μελών για να μην ενταθεί και το φορολογικό άχθος που σηκώνουν στους ώμους τους οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Αυτοί οι νέοι ήδη λοιπόν μπορεί να μειώσουν τις εθνικές συνεισφορές και να μας βγάλουν από την τυραννική ε, ε, αυτή μέγενη του, της επιστροφής για τα κράτη που εποφελούνται και για τα κράτη που συνεισφέρουν. Να ξεφύγουμε λοιπόν από αυτή την ε, μέγενη της δίκαιης επιστροφής των πόρων. Δεσμευόμαστε λοιπόν στο επίπεδο του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου και με τους νέους ε, ίδιους πόρους. Ελπίζω ότι θα εισακουστούμε από το Συμβούλιο, αν και οι πρώτες προβλέψεις δεν είναι εξαιρετικά αισιόδοξε. Όμως έχουμε δεχθεί πιέσεις και εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο ε, και θα πρέπει να ασκήσουμε και εμείς με τη σειρά μας πίεση στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Διότι πρέπει να πάρουμε την κοινή γνώμη με το μέρος μας. Πρέπει η κοινή γνώμη στις χώρες σας ε, και στο ευρωπαϊκό επίπεδο να καταλάβουν το τι ενδιαφέρον έχει αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Μόνο το ευρύτερο κοινό μπορεί να καταλήξει, να πιέσει τους αρχηγούς και των κυβερνήσεων. Τις προκλήσεις και δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την άμυνα, την ψηφιακή ένωση, τις κυβερνοεπιθέσεις, οι πολυεθνικές ε, της ψηφιακής οικονομίας εδράζονται εκτός Ευρώπης, ε, και που οι Ευρωπαίοι ανταγωνίζονται μεταξύ του για να προσκαλέσουν στην επικράτειά του. εδώ βλέπουμε ότι χρειάζεται κοινή ευθύνη και πραγματική αλληλεγγύη. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τι πραγματικέ προκλήσει, φτάνει ο προπολογισμό του 1,2-1,3. Γιατί όχι παραπάνω. Πρέπει να αποδείξουμε όμω ότι Δεν υπάρχει κάποιο δόγμα για τι δημόσιε δαπάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εάν στι εθνικέ σα ε, συζητήσει, στι εθνικέ σα δράσει σα φαίνεται ότι τα εθνικά κράτη στην άσκηση τη εθνική του κυριαρχία σε θέματα άμυνα, ασφαλεία, μετανάστευση ιδίω θέλουν να αντιμετωπίσουν τα αίτια της μετανάστευσης. Αν σας φανεί λοιπόν ότι αυτοί οι πόροι δεν εντοπίζονται σε εθνικό επίπεδο ε, και δεν είναι αρκετά αποτελεσματικοί, αλλά θα είναι πιο αποτελεσματικοί σε ευρωπαϊκό, αυτό μας κάνει να φανταστούμε ότι είναι λογικό οι πόροι που θα προβλέπονταν σε εθνικό επίπεδο να πάνε στον ευρωπαϊκό. Γιατί σε συλλογική χρήση θα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Η αύξηση λοιπόν του ευρωπαϊκού προπολογισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των εθνικών προπολογισμών. Εκεί να γίνουν οι οικονομίες. Η εξυγίανση των δαπανών στην Ευρώπη να επιτρέψει και την πρόοδο της Ευρώπης. Και είναι απαραίτητη και η ευελιξία. Αναφέρθηκε αυτό γιατί χωρί ευελιξία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προσδόκητα γεγονότα και φαινόμενα. Αυτό θα είναι ένα μείζον παράγοντα στι συζητήσει για τον σχεδιασμό του επόμενου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποια είναι η κοινή μα θεώρηση για το μέλλον τη Ευρώπη. Ποια είναι η κοινή μα φιλοδοξία για το μέλλον τη Ευρώπη. Εάν έχουμε ένα κοινό όραμα, μια πραγματική φιλοδοξία, θα πρέπει και να αναλάβουμε τις ανάλογες ευθύνες ως προς τον προπολογισμό και να πείσουμε τα κράτη, τα εθνικά κράτη, ότι για να ε, προετοιμάσουμε το μέλλον για τους συμπολίτε μας, να νιώθουν ασφάλεια, να αισθανθούν εμπιστοσύνη, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Με αυτά τα λόγια σας προτείνω να ξαναδώσουμε ραντεβού στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2018 για την επόμενη διακοινοβουλευτική μας εβδομάδα που θα γίνει και θα οργανωθεί στην Βιέννη, διότι η Προεδρία του Δευτέρου Εξαμήνου του 2018 θα είναι Αυστριακή και εκεί θα μπορέσουμε να ανακεφαλαιώσουμε τα του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου. Εάν θέλετε στις εθνικές σας βουλές, εκεί που είστε μέλη, να οργανώσετε συζήτηση για το ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να μην ξεχνάτε ότι δεσμευόμαστε για την περίοδο 2021-2027 και πραγματικά δεν πρέπει να στοχίσουμε, εάν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Ε, θα κηρύξω λοιπόν τη λήξη αυτής της συνόδου. Σας θυμίζω το ραντεβού που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ την ε, πρόεδρο από την Βουλγαρία που ήταν εξαιρετικά ε, ικανή στο ρόλο της και σας εύχομαι καλή επιστροφή στις χώρες σας και στις εθνικές σας έθνοσυνελεύσεις και βουλές. Γεια σας. Ναι. Ναι.